Uh, uh, λοιπόν, κυρίε και κύριοι, μεγάλη χαρά για μένα να σα ξανακαλωσορίσω σε αυτή την απογευματινή μα συνεδρίαση. Παρακαλώ, καθίστε όλοι και να πω μεγάλο προνόμιο είναι να έχουμε την Επίτροπο κυρία Κουίν ανάμεσά μας φυσικά, Επίτροπος για την Έρευνα και Καινοτομία και είναι ένα άτομο, η κυρία Επίτροπος, που την γνώρισα εγώ και πολλοί ευρωβουλευτές ε, και την μάθαμε από τις τακτικές της επισκέψεις στο σώμα αλλά πιο πολύ θα έλεγα επειδή η δουλειά της για την πολιτική, για την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τόσο μεγάλη σημασία για το μέλλον μας και για μένα είναι ο πυρήνας, το επίκεντρο της ε, Ναυαρχίδας ως πρωτοβουλίας ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση της στρατηγικής του 2020 και να πω ότι είναι το εγχείρημα αυτό, μια και η, ενιαία, η πράξη για την ενιαία αγορά είναι ακριβώς τα θεμέλια αυτών που εσείς θα υλοποιήσετε. Παρ' όλα αυτά παρακολουθήσαμε το έργο σας με ιδιαίτερη θα έλεγα συμπάθεια και ενθουσιασμό και ένα ευρύ φάσμα όσον αφορά το φάσμα δραστηριοτήτων σας όσον αφορά την ενημέρωση αυτή, μια και δεν είναι μόνο για την εκμετάλλευση της καλής έρευνα, αλλά η καλή έρευνα αλλά και η εκμετάλλευση των, των αποτελεσμάτων της και για τα, θέματα της ε, προμήθειας και ε, αγορών και η αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα Χαιρόμαστε που και αυτό το έχετε ως ε, κύρια πρόταση στην στρατηγική για την καινοτομία. Δεν έχει κανείς ε, συχνά την ευκαιρία να καλωσορίζει την Επίτροπο για την Καινοτομία στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, μια και έχετε τόσα πολλά να κάνετε με τις άλλες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Παρακολουθούμε το έργο σας εκ του σύνεγγης, υποστηρίζουμε τις προτάσεις σας και θα το δείτε αυτό μέσα στο πλαίσιο της ε, νομοθεσίας για την ενιαία εσωτερική αγορά. Έχετε τον λόγο, πιέζει ο χρόνος, πρέπει να πάτε σε άλλη Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά οι Ευρωβουλευτές συνάδελφοι θα λάβουν τον λόγο, να διατυπώσουν σίγουρα ερωτήσεις, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε το ρόλο των πολιτικών δημοσίων προμηθειών στην υποστήριξη των στρατηγικών καινοτομία, ιδιαίτερα το βασικό μας στόχο να γίνει η Ένωση Ένωση Καινοτομία. Θέλω να σας δώσω μία εικόνα του ρόλου που οι συνθήκες πλαισίωση, ιδιαίτερα δε οι συγκεκριμένε πολιτικές παίζουν στο πλαίσιο της ε, καινοτομίας ε, όπω υιοθετήθηκαν οι προτάσει αυτέ τον Οκτώβριο. Φέτο η Επιτροπή ανακοίνωσε τους νέους ε, στόχου καινοτομία, που δείχνουν ότι δεν έχουμε προχωρήσει να προφταίνοντα του βασικού ηγέτε στον τομέα, κυρίω στην Ιαπωνία και τη ΣΥΠΑ, ενώ η Κίνα μα προλαβαίνει όλο και περισσότερο. Αυτό πρέπει να είναι ένα ξυπνητήρι για όλου μα και απόδειξη περαιτέρω ότι η Ένωση υποφέρει πάσχει από ένα έλλειμμα καινοτομία. Δεν είναι τυχαίο το ότι είναι πιο καινοτόμοι οι ανταγωνιστέ μα. Είναι διότι έχουν υιοθετήσει στρατηγικέ προσεγγίσει στην καινοτομία που καθοδηγούν όλε τι σχετικέ πολιτικέ και δημοσιονομικέ αποφάσει του. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ηγεσία στην καινοτομία έναντι τη ΕΠΑ και ένα λόγο τη επιτυχία του είναι μια μακρά, ένα μακρό σύστημα υποστήριξη τη καινοτομία που συνδυάζει μέτρα από την πλευρά τη προσφορά με μέτρα ενίσχυση τη διάσταση ζήτηση καινοτομία. με στόχο ιδίω την παροχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, δυνατότητα να προχωρήσουν. Οι ΗΠΑ δαπανούν πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο σε προμήθειε έρευνα και ανάπτυξη, 20 φορέ και περισσότερο από ό,τι η Ένωση. 2 δισεκατομμύρια από αυτό το ποσό πηγαίνει σε μικρομεσαίε επιχειρήσει, σε προγράμματα έρευνα και κοινωνίας με έμφαση στι μικρομεσαιε επιχειρήσει. επιχειρήσεις. Κάποια κράτη-μέλη τη Ένωση έχουν ήδη οθετήσει μια σφαιρική προσέγγιση ε, στην στις προμήθειες έρευνα και ανάπτυξη. Ωστόσο ο κατακαιρματισμός αγοράς σε εθνικό πλαίσιο και η κουλτούρα ε, φόβου του, της διακινδύνευσης στο δημόσιο τομέα εμποδίζουν σημαντικά την προσέγγιση αυτή. Οι δημόσιες συμβάσεις είναι περίπου το, 70%, το 17% της ΑΕΠ, της, του ΑΕΠ της Ένωσης, δηλαδή 2 2-3 εκατομμύρια το χρόνο. Ένα, μια βασική αγορά καινοτομία, ιδίως σε τομείς όπως η υγεία, η οικοδομή, οι μεταφορές και η ενέργεια. Η Ευρώπη λοιπόν έχει τεράστιες ευκαιρίες για να χρησιμοποιήσει την, ε, τις στρατηγικά για να ενισχύσει την κοινοτομία, ενισχύοντας και παροτρύνοντας την δημόσια ζήτηση, η ζήτηση σε τομείς όπου χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες προκλήσεις. Επιπλέον, ε, οι προμήθειες καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών είναι βασική σημασία για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών σε περίοδο λιτότητας. Ένας βασικός στόχος της ε, πολιτικής αυτής στην Ευρώπη, ωστόσο, πρέπει να στρέφει την προσοχή στην καινοτομία. Παρά τις, ε, ε, με, πολλά προβλήματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι συχνά τα κίνητρα μείωσαν τις, δεν έχουν πετύχει τους στόχους, έλλειψη υποδομών και δομών και αποδέσμευση μεταξύ δημοσίων προμηθειών και άλλων πολιτικών στόχων όπως η καινοτομία. Η Ένωση Καινοτομίας έχει συγκεκριμένες προτάσεις για την αύξηση των κονδυλίων για την ε, προμήθεια καινοτομίας, ιδιαίτερα για προϊόντα εμπορικού χαρακτήρα αλλά και, προεμπορικά, ε, και προεμπορικές λύσεις, δηλαδή λύσεις που ακόμα βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας. Η Ένωση κοινωνία ζητά από τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη να, να επιτρέψουν να δημιουργήσουν δομέ και όργανα ε, δημοσίων προμηθειών κοινοτομία που θα παροτρύνουν την καινοτομία και θα υποστηρίξουμε την ανάγκη υποστήριξη καινοτομία στον τομέα στην έκθεση Harbor όπω είχε γίνει το 2006 αλλά και υιοθετώντα την ευρεία στρατηγική του 2007. Οι βασικέ πρωτοβουλίε έθεσαν τρία πιλωτικά σχέδια δημόσιων προμηθειών στον τομέα τη βιώσιμη κατασκευή για τι τοπικέ αρχέ και τα νοσοκομεία και ε, προστα... στην προστασία των, ε, στα προστατευτικά ενδύματα των ε, πυροσβεστών. Αυτή έχει, η προσέγγιση έχει ήδη πετύχει. Ωστόσο, είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, ιδίω παρέχοντα δημοσιονομικά κίνητρα για καινοτομία στην, ε, στις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό συμβαίνει ήδη στα προεμπορικά, στις προεμπορικές συμβάσεις όπου η Γενική Διεύθυνση της Κοινωνίας της Πληροφορίας έχει προχωρήσει στην υποστήριξη Ευρωπαίων ε, αναδόχων σε πράξεις ε, ε, προμήθειας. Ήδη υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του, του προγράμματος πλαισίου 7 για να υπάρξει δημόσια κρατική υποστήριξη των προεμπορικών της καινοτομίας στις προεμπορικές ε, συμβάσεις. Η, ομάδα, η Συρική ομάδα θα εξασφαλίσει το ότι αυτά τα μέτρα θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση πανευρωπαϊκών μέτρων καινοτομία. Με βάση μια μελέτη σκοπιμότητα που προχωρεί αυτή τη στιγμή, ο στόχο μα είναι να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα υποστήριξη τη προμήθεια στην καινοτομία σε ε, ευρεία κλίμακα ούτω ώστε να υπάρχει προεμπορική καινοτομία για μελλοντικά έργα. Ο Αντιπρόεδρος κ. Σταγιάννη θα ξεκινήσει ένα πιλωτικό σχήμα 15 εκατομμυρίων ευρώ φέτος το καλοκαίρι για την προμήθεια καινοτομία και προεμπορική καινοτομία, ούτω ώστε να παράσχει το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για αυτό το μελλοντικό ε, ευρωπαϊκό σχέδιο. Πολλέ περιφέρειε έχουν προχωρήσει σε τέτοια μέτρα. Άλλε περιφέρειε προχωρούν ή προσαρμόζουν υφιστάμενα προγράμματα. Τα καλωσορίζουμε και τα υποστηρίζουμε. Θέλω να στραφώ τώρα στην κύρια εικόνα, στη γενική εικόνα της καινοτομίας. Η κατάσταση, πρόεδρε, σήμερα συμβαίνει μια, σε μια, η συζήτηση συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Ε, την Πέμπτη θα συναντηθούν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και συζητήσουν μεταξύ άλλων και την καινοτομία. Τι θα αποφασίσουν. Πρώτον, όπω οι ανταγωνιστέ μα και κάποια κράτη-μέλη κάνουν ήδη, η Ένωση πρέπει να υιοθετήσει μια στρατηγική προσέγγιση ενίσχυση και παρότριση τη καινοτομία βάσει των βασικών, ε, σχε, των βασικών θέσεων τη ενό καινοτομία, όντα καλύτερη, ταχύτερη και προσφέροντας καλύτερες ιδέες στην αγορά. Παρά, έχουμε παράσχει μια σειρά προτάσεων για την επίτευξη κάτι τέτοιου, συμπεριλαμβανομένων και των στρατηγική χρήση των δημόσιων προμηθειών. Δεύτερον, σε μια φάση δημοσιονομικής λιτότητας πρέπει να προωθήσουμε έξυπνη ε, δημοσιονομική παγίωση προσφέροντας επενδύσεις όσο καλύτερα γίνεται στην παιδεία, την έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την έξυπνη υποδομή καθώς και φιλόδοξες μορφές εθνικών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας. Τομείς από όπου εξαρτώνται πολλές θέσεις εργασίας, κινητοποιώντας η κινητοποίηση δημοσίων προμηθειών για την καινοτομία είναι μοναδική για την, στον τομέα αυτό, προσφέροντας ευκολότερα και γρηγορότερα καρπού σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και με ευκολότερες ε, αποδόσεις στις επενδύσεις που κάνουμε οι συμβάσεις καινοτόμε λύσεις σημαίνει ότι ε, μέσω πρόθεσμα η κοστοποτελεσματικότητα μέσω ε, εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί και να καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, οι δημόσιες προμήθειες μπορεί να δώσουν καλύτερη απόδοση στα χρήματα των φορολογούμενων. Τρίτον, χρειαζόμαστε εξυπνότερα ε, εξυπνότερη πλαισίωση, να υιοθετήσουμε ένα περιβάλλον με μεγαλύτερη να πάω λίγο πιο αργά, λέει η ομιλήτρια. Τρίτε, να υιοθετήσουμε ένα πλαίσιο που θα οδηγεί ευκολότερα στην κοινοτομία και θα, παρέ, και θα έχει καλύτερη θέση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό ούτως ώστε να προσελκύσει και να κρατήσει και την ιδιωτική επένδυση και το ταλέντο. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε το πλαίσιο σε τομείς όπως η πνευματική ιδιοκτησία, διπλώματα ευρεσιτεχνία, πρόσβαση σε κεφάλαιο διακινδύνευσης, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης θα εξετάσουμε τις οδηγίες της Ένωσης σχετικά, χρησιμοποιώντας την την ε, πρόσφατη αξιολόγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αγορά, Εσωτερικής Αγοράς των Οδηγιών του 2004 για να εξυγχρονίσουμε το κείμενο χρειάζεται, βοηθώντας την προώθηση της καινοτομία μέσω της διαδικασίας ε, ε, δημοσίων προμηθειών. Ξέρω ότι και εσείς είστε πεπισμένοι για την ανάγκη βελτίωσης των προδιαγραφών και της τυποποίησης. Η Επιτροπή την Άνοιξη θα υποβάλει μια ανακοίνωση και μια νομοθετική πρόταση για την τυποποίηση, ούτω ώστε να επιταχύνει και να ξυγχρονίσει την θέσπιση προτύπων για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και την νίκηση της καινοτομία στην ταχεία εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά. Σε συνδυασμό θα γίνει αυτό με ένα παγκόσμιο πολιετές, με ένα πολιετές πρόγραμμα που θα ενσωματώνει τα πρότυπα στα προϊόντα έρευνας και ανάπτυξης στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Τέταρτον, πρέπει να διερευνήσουμε όσο καλύτερα γίνεται την θέμενη αξία των δράσεων της Ένωσης και να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας όπως ε, η αντιμετώπιση τη αλλαγή του κλίματος χρησιμοποιώντας τους σπάνιου πόρου πιο αποτελεσματικό και να φροντίζουμε περισσότερο τους ηλικιωμένου μας. Θα ξεκινήσουμε μια μικρά, ένα μικρό αριθμό εταιρικών, εταιρικών σχέσεων στην καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με συγκεκριμένου στόχου. Ένα βασικό κριτήριο επιλογής για τα αυτά θα είναι να υπάρξει δυναμικό στην αγορά για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες και να υπάρχουν ευρωπαϊκές εταιρείες που θα είναι πρωτοπόροι στον τομέα. Η εταιρική αυτή σχέση θα φέρει στην, στον ίδιο χώρο όλους τους εμπλεκόμενους, συνδυάζοντας μέτρα προσφοράς και μέτρα ζήτησης, αλλά και, και πρότυπα και νομοθετική ρύθμιση. Τα κράτη-μέλη θα εμπλέκονται σε αυτές τις εταιρικέ σχέσεις και θα μπορούν να κινητοποιήσουν την ζήτηση μέσω στρατηγικών προγραμμάτων καινοτομία, για παράδειγμα και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο υποστήριξε αυτή την ε, πρωτοβουλία με το ψήφισμά του στις 11 Οκτωβρίου. Ε, μια πιλωτική εταιρική σχέση έχει ήδη ξεκινήσει και ο στόχος είναι το 2020 να επεκτείνει την μέση υγεία, η υγιεινή ζωή του Ευρωπαίου κατά δύο έτη. Το Κοινοβούλιο θα εμπλακεί πλήρως και ε, στην πιλωτική διάσταση και στην πλήρη εφαρμογή της διάταξης. Αυτές είναι οι τρεις πρώτες προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας ένωσης καινοτομία. Αλλά υπάρχει και άλλη μία. Το η βάση επί της οποίας βασίζονται όλες οι δράσεις μας. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πρέπει να αναλάβουν ευθύνη για την εφαρμογή της Ένωσης ε, Καινοτομίας και να παρακολουθούν τακτικά την πρόοδο. Βεβαίως, δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Υπουργών που θα το κάνει αυτό, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει σημαντικό ρόλο να παίξει και ειδικά η Επιτροπή σας που έχει σημαντικές ευθύνες για ζητήματα δημοσίων προμηθειών και άλλα. Βεβαίως, έχετε και ένα βασικό ρόλο στην σύνταξη της γνώμης του Κοινοβουλίου για την Ένωση της Καινοτομίας. Είμαι πεπισμένη πως η συγκεντριά σας θα κάνει πάρα πολύ καλό έργο. Και θα σα ζητούσα να κάνετε ακόμη περισσότερα εάν θέλουμε να επιτύχουμε ή να ξεπεράσουμε τον στόχο των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ ανά έτος. Και άρα χρειαζόμαστε την εμπλοκή όλων των δημοσίων αρχών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών. Γνωρίζω πως το ζήτημα των δημοσίων προμηθειών απασχολεί πάρα πολύ τον κύριο Χάρμπορ και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, οπότε θα σας ζητούσα να χρησιμοποιήσετε την επιρροή σας, συναδέλφους σας στα κράτη-μέλη, για να τους ενθαρρύνετε να αναλάβουν αυτή την πρόκληση και να ανταποκριθούμε στους κοινούς μας στόχους για, την... για τις προμήθειες στην καινοτομία. Πάρα πολλά μπορούμε να επιτύχουμε και βεβαίως με υποστηρικτές σε όλο το πολιτικό φάσμα είμαι σίγουρη ότι θα επιτύχουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Νομίζω πως όλοι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το ότι οι προμήθειες για την καινοτομία επιτέλους βρίσκονται στην κορυφή των ε, θεμάτων πλέον, γιατί ήταν κάτι που ζητούσαμε εδώ και χρόνια. Λοιπόν, έχουμε πολλού συναδέλφου. Ο κ. Τριανταφυλλίδη είναι ο εισηγητή. Το πότε θα έχει πρώτο τον λόγο. Η κυρία Ρούλη είναι η εισηγήτρια για τι δημόσιε προμήθειε. Οπότε θα λάβει και εκείνη τον λόγο. Ακούσουμε λοιπόν πρώτα αυτού του δύο και μετά Schwab, Στάιλερ και Βάιλερ μέχρι στιγμή και Κορέα Campos. 25 λεπτά έχουμε συνάδελφοι γιατί μετά έχουμε την ψηφοφορία και εσείς πρέπει να πάτε βέβαια σε άλλη επιτροπή. Οπότε θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομοι, να μιλήσουμε τρεις-τρεις. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης, η κυρία Ριούλα και ο κύριος Σβάμπ. Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την Επίτροπο για την παρουσίασή της. Κατά την άποψή μας, οι μεγαλύτερες αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή που υποσκάπτουν τη δυνατότητα περαιτέρω διεισδυτικότητα σε νέες αγορές παγκόσμια αφορούν πρώτον ανεπαρκείς επενδύσεις στο γνωστικό της κεφάλαιο. Όπως είπε και η Επίτροπος, άλλες χώρες όπως η ΙΠΑ και η Ιαπωνία πραγματοποιούν μεγαλύτερες επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να καλύπτει πολύ γρήγορα τη διαφορά. Δεύτερον, μη ικανοποιητικέ συνθήκες πλαισίου από τις δυσκολίες στην εξέβρεση χρηματοδότησης. Πρόκειται για πολύ σοβαρό μειονέκτημα αφού οι εταιρείε μπορούν να επιλέξουν να επενδύσουν και να πραγματοποιήσουν έρευνα σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Και τρίτον, καταγερματισμός προσπαθειών και δαπανηρή επανάληψη εργασιών. Συνεπώς, κατά την αντίληψή μας, οι άξονες δράση μας θα πρέπει να επικεντρωθούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να διευκολύνουμε τις διαδικασίες χρηματοδότησης ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υπερβούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διαδικασία ανάληψης χρηματοδότησης και ταυτόχρονα να βρούμε τρόπους ενθάρρυνσης της κρίσης καινοτόμων λύσεων. Άρα καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση ώστε να μην αποθούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικονομικά προσιτοί. Στο δημόσιο τομέα η καινοτομία θα πρέπει να σταθεί αρρωγός στην προσπάθεια διευκόλυνσης των διοικητικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και στη μείωση της γραφειοκρατίας και της δισκαμψίας του δημόσιου τομέα με την εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων. Οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένα μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να εισαγάγουν στη διαδικασία των δημόσιων συμβάσεων τον τομέα της καινοτομίας. Τελειώνω. Επιπροσθέτω, η υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τι προεμπορικέ συμβάσει, οι οποίε επιλύουν ζητήματα που αδυνατεί να καλύψει η αγορά ή οι λύσει που προτείνονται είναι ασύμφορε. Η μέθοδο των προεμπορικών συμβάσεων αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη αυτών των προγραμμάτων και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στου πολίτε. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Τριανταφυλλίδη. Σας έδωσα χρόνο γιατί είστε και συγητή, οπότε ξέρει η κυρία Γκέγεν Κουίν τι την περιμένει. Αν οι υπόλοιποι συνάδελφοι μπορούν να είναι λίγο πιο σύντομοι, θα ήταν καλό. Κύριε Ρούλα. και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Όταν ε, είδα το θέμα των δημοσίων προμηθειών παρατήρησα πως πολλές τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν ξέρουν πολλά πράγματα για τα νομικά αυτά μέσα, π.χ. για τα προσύμφωνα αυτά, τις ε, προεμπορικές ε, συμφωνίες, δεν έχουν πληροφορίες. Οπότε σημαντικό είναι να οδηγηθούμε σε καλύτερη πληροφόρηση και αυτό το οποίο είπατε είναι κατακαιρματισμένη η αγορά Οπότε το ερώτημα είναι εάν υπάρχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για καλύτερη συνεργασία των ε, δημοσίων προμηθειών, γιατί εκεί πέρα υπάρχει πολύ δυναμικό και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως είναι δυνατόν να γίνουν τέτοιες συνεργασίες χωρίς να οδηγηθούμε σε καρτέλ. Ξέρω πως είναι δυνατόν, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες. Δεύτερο ερώτημα, στην πράσινη στις πράσινες προμήθειες υπάρχει μια πολύ επιτυχημένη ΜΚΟ η Ίκλη που εργάζεται εκεί πέρα και οργανώνει σεμινάρια και βοηθάει τις, ε, τους Δήμους να πάνε προς τις πράσινες προμήθειες. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια καινοτομία, συνεργασία με ΜΚΟ για να έχουμε καλύτερη πληροφόρηση. Και υπήρχε και η αρχή του Frontrunner, δηλαδή να υπάρχει ένας ανταγωνισμός για να δούμε ποιο κράτος θα τα καταφέρει καλύτερα και να υπάρχει έτσι και ένα κίνητρο να κάνουν τα κράτη περισσότερα. Αυτή είναι η μέθοδο, δηλαδή να έχουμε ένα ΜΚΟ συνομιλητή και να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη υπό μορφή έτσι, ανταγωνισμού. Αυτέ είναι οι παρατηρήσεις που έχω να κάνω. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε και από πλευρά μου φυσικά είναι μεγάλη χαρά πρέπει να πω ότι είσαστε παρούσα στην κοινοβουλευτική μας Επιτροπή και μας αναφέρετε αυτό το σημαντικό θέμα. Καταρχήν πρέπει να δούμε πιο εξειδικευμένα το θέμα στην έκθεση του κυρίου Τριανταφυλλίδη και πώς η καινοτομία μέσα στο πλαίσιο των συμβάσεων θα καθορίζεται. Είναι σαφές ότι θα έχουμε νέα νέες λύσεις θελκτικές και λειτουργικές για τους πολίτες αλλά δεν πρέπει με πρόσχημα την καινοτομία να δημιουργηθούν εμπόδια για τις συμβάσεις ε, και προμήθειες. Και γι' αυτό θα ήθελα να προσθέσω τη φωνή μου σε αυτά που είπε η κυρία Ρούιλε σε σχέση με τους φορείς. Ε, θα πρέπει να δούμε ότι το δυναμικό της αγοράς μόνο σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος προσφοράς ε, μπορεί να λειτουργήσει. Και επιμέρους ίσως θα είναι αναγκαίο σε σχέση με επιμέρους φορείς τις ε, συγκρούσεις ε, ή τις, ε, τα θέματα να τα δεχθούμε μέσα σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού. Πρέπει όμως και περισσότερα κονδύλια να μπορέσουν να επενδυθούν στην καινοτομία και την έρευνα. Διαφορετικά από ό,τι εσείς ε, προηγούμενα αναφέρατε ή αναφέρθηκε πιο πριν για την Κίνα και της είπα ότι δεν χρειάζεται να τις φοβόμαστε, ότι δεν είναι αρνητική η θέση μας ως Ευρώπης, αλλά σε σχέση και με το θεματολόγιο 2020 όπου γίνεται λόγος ε, για καινοτομία και ότι τα όρια της καινοτομίας θέλουμε να τα διευρύνουμε και δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εθνική ιδιομορφία γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ε, Κύριε Επίτροπε, θα θέλετε να απαντήσετε σε αυτά πρώτα τα ερωτήματα και μετά θα ακούσουμε την κυρία Στάιλερ, τον κύριο Βάιλερ και Κορία Ντεκάμπους. Και κλείνει ο κατάλογος ομιλητών. Κυρία Επίτροπε, Πράγματι, κάθε ένας από τους τρεις ε, βουλευτές, δεν, ο εισηγητής θα με συγχωρήσει, δεν θα προσπαθήσω καν να προφέρω το όνομά του, γιατί πραγματικά θα κάνω λάθος και θα τον προσβάλλω. Όλα τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν από τους τρεις ομιλητές βεβαίω ε, απασχολούν πάρα πολύ εμένα και τις υπηρεσίες μου. Δηλαδή πώς βλέπουμε τον εαυτό μας στον τομέα αυτών, πώς στεκόμαστε σε σχέση με τους άλλους και νομίζω πως ως διαγνωστικό μέσο αυτός ο πίνακας βαθμολογίας που έχουμε είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός για να δούμε πώς στεκόμαστε όχι μόνο σχέση ο ένας με τον άλλον αλλά με τη ΣΥΠΑ, Κίνα και Ιαπωνία. Και όταν βλέπουμε τις επενδύσεις που γίνονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτών δεν ε, είμαστε τόσο επιτυχείς πολύ συχνά. Προσπαθήσαμε λοιπόν όταν στείναμε αυτή την πολιτική για την Ένωση της Κοινοτομίας να δούμε πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Και κοιτάξτε εγώ μόλις είχα επιστρέψει από τη ΣΥΠΑ, όπως ξέρει ο Μάλκομ, όπου είχα συζητήσει όλη αυτή την πολιτική ε, SBIR ε, που εφαρμόζει ο πρόεδρος Ομπάμα και το πώς, το πώς ε, το εφαρμόζουμε τον αρμόδιο υπουργό. Και βεβαίως με το να θέτουμε το πλαίσιο για να επενδύσουν τα κράτη-μέλη σε καινοτόμες ε, δημόσιες προμήθειες ή προεμπορικές συμφωνίες. Όταν είπαμε για 10 δισεκατομμύρια όλοι μας είπαν πως ήμασταν πάρα πολύ συντηρητικοί και έπρεπε να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι. Εγώ θεωρούσαμε το ότι με το να είμαστε λίγο συντηρητική θα υπήρχε μια όθηση στα κρατημέλη για να πάνε ακόμη παραπέρα από αυτά τα οποία τους είχαμε ζητήσει. Είναι ενδιαφέρον. Έχουμε παραδείγματα, ξέρετε, παραδείγματα εντός της Ένωσης όπου έχει ακολουθηθεί ένας δρόμος ανάλογος με το SBIR. Είναι όμως ενδιαφέρον πως από πλευράς αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων να εξετάσει ο καθένας το τι μπορεί να γίνει στον τομέα υποστήριξης για προεμπορικέ συμφωνίες και δημόσιες καινοτόμε προμήθειες. Βεβαίω αυτά τα 10 δισεκατομμύρια είναι μια φιλοδοξία, είναι απλά για να ξεκινήσει η όλη υπόθεση. Να φτάσουμε έτσι σε ένα σημείο μετά από το οποίο θα αρχίσουν να υπάρχουν εξελίξεις. Δεν είναι δηλαδή ε, μια υποχρέωση είναι ένας στόχος και ε, είναι αυτό το οποίο θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε από πλευρά κομισιών. Επίσης αναφέρεται σε συγκεκριμένες δημόσιες προμήθειες που βρίσκονται σε μια προεμπορική φάση για αγορές παραδείγματος χάρη νέας τεχνολογίας ή καινοτομιών ως μέρος ε, της εφαρμογής των ευρωπαϊκών συνεργασιών καινοτομίας. Βεβαίως εμείς ως Κομισιόν θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία του μηχανισμού στήριξης και βεβαίως μέσω των εταιρικών αυτών σχέσεων καινοτομία, αλλά πρέπει να θυμόμαστε πως 17% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ προέρχεται από τις δημόσιες προμήθειες και αυτός είναι ένας τομέας που πρέπει να επιδείξει καινοτομία. Π.χ. κοινέ προμήθειες χωρών, περιφερειών, διασυνοριακά. Να δούμε πώς μπορούν να συνεργαστούν και τίποτα δεν τους εμποδίζει να συνεργαστούν. Και ήδη, παραδείγματο χάρη όταν ε, μιλάμε για τοπικές αρχές, περιφέρειες, ε, το πώς μπορούν να συνεργαστούν, δεν τους εμποδίζει τίποτα να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί ήδη αυτό γίνεται εντός του, της χρηματοδότησης του προγράμματος πλαισίου 7. Δεν νομίζω πως θα ήταν σωστό η Κομισιόν να νομοθετήσει αλλά νομίζω πως ε, είναι κάτι το φιλόδοξο και ελπίζω, όπως είπα, να αλλάξει την ισορροπία προς σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά τώρα τον ορισμό της καινοτομίας, ο κύριος Σφάπ το ανέφερε, αυτό εξαρτάται και από το πώς οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να ενθαρρυνθούν για να συνεργαστούν. Και μην ξεχνάμε πώς θα ξεκινήσουμε την άλλη εβδομάδα μια μεγάλη διαδικασία διαβούλευσης ε, για το επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την κοινοτική έρευνα και καινοτομία και αυτό θα γίνει με τρόπο καινοτόμο και συνολικό που θα ξεκινήσει από τις περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι ευκαιρία για τον κόσμο να αντιληφθεί το πώς μπορεί να συνεργαστεί ο ένας με τον Πράσινε προμήθειες, ναι, πολύ σημαντικές βεβαίω. Είναι ένα τομέα που μας έχει απασχολήσει πολύ. Θέλουμε να συνεργαστούμε με τους πάντες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. ΜΚΟ, τοπική αυτοδιοίκηση, κυβερνήσεις κρατών μελών. Πρέπει να συνεργαστούμε, να του εμπλέξουμε στο σύστημα ή να προωθήσουμε αυτό το θέμα των δημοσίων προμηθειών ως ένα τομέα στον οποίο μπορούμε να κερδίσουμε πολλά και όπου, παραδείγματο χάρη, οι Ηνωμένε Πολιτείες ζηλεύουν τις αρμοδιότητες ε, δημοσίων προμηθειών που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε που προχωρήσατε τη συζήτηση. Οι τελευταίοι τρεις ομιλητές και θα ήθελα να τους παρακαλέσω να είναι σύντομοι η κυρία Στάιλερ, η κυρία Βάιλερ και ο κύριος Κορέα Ντεκάμπος. Κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας έχουμε σήμερα στην Επιτροπή. Μιλήσατε για το τι γίνεται στις Ηνωμένες Διαπιστώσα σήμερα ότι η έκθεση του Ομπάμα για, τη, για τις επενδύσεις λέει, ε, παρέχει τη δυνατότητα ε, να εκπέσεις τις επενδύσεις στην καινοτομία για να ξαναφέρνεις χρήματα στο σύστημα. Εμείς πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια πολιτική. Εμείς έχουμε την προοπτική της Ευρώπης 2020, την ψηφιακή ε, ε, και την ψηφιακή ημερήσια διάταξη. Εσείς θεωρείτε ότι η ψηφιακή ημερήσια διάταξη και η ημερήσια διάταξη για την καινοτομία κολλάνε μεταξύ τους. Επίση, πώ μπορούμε να συνδέσουμε αυτή την πολιτική με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η κυρία Βάιλερ. Και εγώ θα είμαι σύντομη. Μια στιγμή το τσάι παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επανέλθω στην απάντησή σας στην ερώτηση της κυρίας Ροϊλέ για τη συνεργασία. Φυσικά είναι σαφές ότι με όλους θέλουμε να συνεργαστούμε και σίγουρα με σθένος θα το κάνουμε. Το θέμα, το ερώτημα είναι αν με αυτόν τον τρόπο επιλέγεται μία ΜΚΟ που θα είναι υπεύθυνη για πράσινη πολιτική, για τις πράσινες ε, προμήθειες ή και για την καινοτομία. Αν από πλευρά σας ενεργά θα επιλέξετε, θα συμμετάσχετε σε αυτήν την επιλογή, γιατί διαφορετικά πέντε χρόνια θα κρατήσει πάλι όλο αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είπατε ότι δεν θέλετε να νομοθετήσετε ε, τότε σίγουρα εκινείται από την αφετηρία ότι όχι μόνο δεν επαρκεί μια ανακοίνωση της Επιτροπής, αλλά πρέπει να κάνετε πιλωτικά προγράμματα, κυρίως το 7ο και 8ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Μπορείτε να μας αναφέρετε ήδη ένα πρόγραμμα πιλότο που να λειτουργήσε με καινοτόμες πτυχές όπως τα φαντάζεστε εσείς ή κάτι άλλο όπως εσείς στοχεύετε να πορευτείτε για την καινοτομία και τα πρότυπα, τα πιλωτικά τέτοια προγράμματα. Έχετε κάτι να μας πείτε. Thank you very much, uh, ο καθηγητής Κορέα Ντεκάμπος, ευχαριστώ Επίτροπε. Είναι χαρά να σας έχουμε Επίτροπε εδώ ανάμεσά μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής η φιλοδοξία σας. Μπορείτε να μας πείτε, θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε, στοχεύει στο να δημιουργηθεί μια ενιαία εσωτερική αγορά για την καινοτομία. Είναι εφικτό να έχουμε μια ενιαία εσωτερική αγορά για την καινοτομία και τα βήματα που θα γίνουν θα είναι για να δημιουργηθεί αυτή η ενιαία εσωτερική αγορά ή όχι. Σε σχέση με τα, τις συμβάσεις και τα 10 δισεκατομμύρια που θα είναι αναγκαίο για την, αναγκαία για την καινοτομία, τα συγκρίνουμε βέβαια με τα 50 δισεκατομμύρια των Βορειοαμερικανών, των ΗΠΑ. Συμφωνούμε με τα θέματα ανταγωνισμού και για τα θέματα ανταγωνισμού όσον αφορά την διασφάλιση αυτών των κονδυλίων. Όμως έχουμε και τις αναδυόμενες οικονομίες των χωρών όπως η Ινδία και η Κίνα που έχουν διαμετρικά αντίθετες ε, ιδεολογίες και μεθοδολογίες από εμάς για τον ανταγωνισμό. Η ερώτηση που θέτω, σκέφτεται να συνδυάσετε κάποια μεθοδολογία για τα θέματα ανταγωνισμού που θα είναι ενεργής, ε, ενεργού χαρακτήρα ή όχι. Ευχαριστώ. Η θα απαντήσει. Um, Για την τελευταία ερώτηση να απαντήσω πρώτα. Βεβαίως, αυτό θέλουμε να κάνουμε, να έχουμε ανανέωση της ενιαίας αγοράς. Αυτό το είπαμε εξ αρχής, πιστεύουμε ότι αυτή είναι η σωστή πορεία. Συχνά ανέφερα και στο Κοινοβούλιο και εκτός ότι ανάλογα με το πώς η Ένωση αντιμετωπίσει την καινοτομία θα σημαίνει κατά πόσον ανοίγουμε ή κλείνουμε σε σαν επιχείρηση. Υπάρχει μια, μια ανάγκη καινοτομίας, έκτακτη ανάγκη καινοτομίας. Το συζητούμε επί ένα χρόνο, το εξηγούμε στα κράτη-μέλη, στα Συμβούλια Ανταγωνισμού, στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Ήτρε, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Το αποκορύφωμα όλων αυτών είναι ότι για πρώτη φορά οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων την Πέμπτη θα κάτσουν να συζητήσουν τα θέματα της καινοτομίας και της ένωσης καινοτομίας στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν ένα παράθυρο ευκαιρία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διότι μπορεί να αργήσει να ξανανοίξει. Επίσης έχουμε μια κατάσταση όπου σε παγκόσμιο επίπεδο η δήλωση του Ομπάμα για, το, για την κατάσταση της Ένωσης περιλαμβάνει σαν κλειδί την καινοτομία. Δεν το λέμε λοιπόν μόνο εμείς, το λένε οι ΙΠΑ. Και πάντα κοιτάμε προς τη Δύση. Δείτε όμως και την Ανατολή. Μας έχει φτάσει πίσω από το λαιμό μας αυτή τη στιγμή η Κίνα. Γι' αυτό το λόγο πιεζόμαστε και γι' αυτό μιλάμε για το σύνθημα Ένωση Καινοτομίας. Ο κύριος Ντε πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο από τον πίνακα επίδοσης ε, στην κοινοτομία του κράτους που γνωρίζει καλύτερα. Τώρα, η ΜΚΟ. Πολύ σημαντική συνεργασία με ΜΚΟ. Οπουδήποτε βρούμε οργανώσεις, ανθρώπους, τοπική αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ ε, που μπαίνουν σε προμήθειες είτε στον πράσινο τομέα είτε αλλού πρέπει να μετάσχουν. Χρειαζόμαστε να μετάσχουν. Ήδη, όπως ξέρετε, μετέχουν στα, σε κονσόρτια του προγράμματος πλαισίου 7. Δεν τους εμποδίζει κάτι τέτοιο. Θέλουμε να το προωθήσουμε, θέλουμε να πουλήσουμε το αντίστοιχο μήνυμα και χρειαζόμαστε όλους σας να δώσετε στα κράτη-μέλη, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και κυβερνήσεις αυτό που θέλουμε να περάσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που μπορείτε να περάσετε με εξαιρετικά αποτελεσματικότερο τρόπο που μπορούμε να, ε, μπορείτε να περάσετε στους πολίτες σας. Η χρήση κονδυλίων της καινοτομίας με έξυπνο τρόπο είναι σημαντικό. Η, καινο, η, ψηφιακή ατζέντα και η ατζέντα ε, καινοτομίας είναι συμπληρωματικές. Δείτε ωστόσο την κατάσταση. Ε, η πιλωτική εταιρική σχέση είναι μπροστά. Παίζουν η ψηφιακή ατζέντα, είναι πολύ σημαντική για την Ένωση Καινοτομία και για τη συνεργασία. Όπω σα είπα, χρειαζόμαστε και πιλωτικά έργα. Όταν μιλούσα στο, στην αρχή, είπα ότι είχαμε προσυμβατική ε, προσυμβατικές ρυθμίσεις, ρυθμίσεις για τις προσυμβατικές συμβάσεις και προμήθειες. Έχουμε μηχανισμό ο πρώτος μηχανισμός υποστήριξη από πλευρά τη Επιτροπής είναι διαθέσιμος μέσω του προγράμματος εργασία ICT, του 7ου προγράμματος Πελσίου, για να δώσουμε ε, υποστήριξη για την κοινή εφαρμογή των προ-συμβατικών ε, ε, προμηθειών. Βεβαίως αυτό είναι το ξεκίνημα. Τώρα προχωρούμε με έναν οδικό χάρτη για να ετοιμάσουμε πολιτικές που θα ξεκινήσουν την άλλη εβδομάδα με αυτή την σημαντική εμπλοκή του κοινού σε όλες τις ε, χώρες της Ένωσης και με, για να δούμε πώς θα είναι το μελλοντικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Καταρχάς, διότι δεχθήκατε να έρθετε εδώ, διότι παρουσιάσατε με σαφή τρόπο τις ιδέες σας για το μέλλον. Θα έλεγα, θα έπρεπε να είχα πει αυτό από την αρχή, ότι αυτό είναι κομμάτι της ε, στρατηγική συνεργασία μας με την Επιτροπή, αλλά το αναφέρετε κι εσείς. Έπρεπε να είχα αναφέρει και τα πρότυπα. Είναι ένα τομέα που έχει μεγάλη άλληλο επίδραση. Σας ευχαριστώ εκ νέου που ήρθατε και ευχαριστώ που αντιμετωπίσατε ε, και απαντήσετε σε όλε τι ερωτήσει μα. Θα ξεκινήσουμε ψηφοφορίε τώρα, ξέρετε κάτι πολύ συγκλονιστικό πάντα. Θα πάτε σε άλλη επιτροπή, αλλά θα ήθελα να σας δώσω και ένα δωράκι από την επιτροπή μας. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα support group της Ιρλανδίας πολύ ισχυρό. Ξέρετε ότι σήμερα είναι η μέρα της Αγίας Bridget. Πολύ αυτό. Σας δίνουμε λοιπόν έναν σταυρό της Αγίας. Φαντάζομαι μόνο εμείς θα σας δώσουμε τέτοιο δώρο σήμερα. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Uh, λοιπόν κυρίες και κύριοι uh, could I, um, we now have a long... Έχουμε τώρα μακρά συνεδρίαση με ψηφοφορίες. Καθίστε παρακαλώ όλοι σας. Αν όλοι μπορούν να καθίσουν θα ήταν καλό. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Uh, we will θα χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες για την ψηφοφορία, μια και έχουμε πολλές ψηφοφορίες. Διασφαλίστε ότι έχετε τις κάρτες σας όλοι. Θα έχουμε την εναρκτήρια ψηφοφορία για να ελέγξουμε πώς είναι παρόντες και τι γίνεται. Είναι όλοι παρόντες τώρα εδώ. Uh, Λίγη ησυχία παρακαλώ. Right. Λοιπόν, θα ελέγξουμε με μια ηλεκτρονική ψηφοφορία το σύστημα πριν ξεκινήσουμε επίσημα με τις ψηφοφορίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Καλό τα μέλη του ΕΛΚ να ψηφίσουν τώρα. Τα μέλη του ΕΛΚ παρακαλώ ψηφίστε τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία για το ΕΛΚ. Ψηφίσατε όλοι, είναι όλοι παρόντες. Όχι. Οκτώ καταφέρατε και βρήκατε. Έρχονται κι άλλοι. What? All right. Λοιπόν, πέρα ψηφοφορία για τα μέλη του ΕΛΚΑ. Έχουν αρκετή δουλειά μέχρι να τους φέρουν όλους, στην αίθουσα. Άρχεται η ψηφοφορία για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Άρχεται. Είναι σίγουρα παραπάνω από έξι μέλη των σοσιαλδημοκρατών εδώ. Βλέπω αρκετούς ήδη. Σοσιαλδημοκράτες παρακαλώ να συμμετάχουν στην ψηφοφορία. Οκτώ Λοιπόν, περισσότεροι θα έρθουν. Έρχονται, εντάξει. Βλέπουμε του υπόλοιπου. Τρεις φιλελεύθερου, δύο πράσινους βλέπω. Λοιπόν, οι σοσιαλδημοκράτε είναι η μόνη δύναμη, η μόνη κομματική ομάδα που έχει τον πλήρη αριθμό. Μέχρι στιγμή η μικρή είναι εντάξει. Λοιπόν, προχωρούμε και ψηφίζουμε πρώτα την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας ε, Σάλε Μόσα για την οδηγία για την ασφάλεια και την εποπτεία των αγορών, ασφάλεια προϊόντων. Η συγγήτρια θα ήθελε να πει δύο λόγια πριν από την ψηφοφορία να μας εισαγάγεται στο θέμα της ψηφοφορίας, παρακαλώ. Θα σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι θα είμαι σύντομη γνωρίζω ότι έχουμε μακρά ψηφοφορία ενώπιόν μας, όχι τόσο για τη δική μου την έκθεση, αλλά ιδιαίτερα για την έκθεση που ακολουθεί την δική μου μετά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οκτώ συμβιβαστικές τροπολογίες έχουμε ενώπιόν μας για την έκθεση, για την ασφάλεια προϊόντων, και αυτό τι σημαίνει με άλλα λόγια. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια έκθεση που με μεγάλη υποστήριξη και μεγάλη συνένεση πρέπει να πετύχουμε στην έκθεσή μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αν μια έκθεση πρέπει να είναι ένα σαφές μήνυμα αυτό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μια επανεξέταση της οδηγίας για την ασφάλεια είναι εκείνο που χρειαζόμαστε. Όμως και πρέπει να ενισχυθεί και η εποπτεία, η επόπτευση της αγοράς, διότι δεν λειτουργούν τα πράγματα αυτή τη στιγμή αρκετά καλά και θεωρούμε, συνενούμε συνενετικά ως ε, ομάδες ε, πέρα από κομματικά όρια. Χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό σύστημα εποπτείας των αγορών και αυτό ζητάμε κιόλα εξάλλου με αυτή την έκθεση. Ελπίζω όμως ότι όλα αυτά θα έχουν θετική έκβαση και θα γίνουν δεκτά. Και θέλω να δραχθώ της ευκαιρίας ώστε να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία σε σχέση με τις συμβαστικές τροπολογίες και για την εκπόνηση της έκθεσης γενικότερα. Δεν είναι απλά τα πράγματα όταν έχουμε διαφορετικές και θέσεις να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό. Αυτό σημαίνει ότι αφενός η ασφάλεια για τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά ενισχύεται. Από την άλλη όμως πλευρά και για τις επιχειρήσεις διευκολύνονται τα πράγματα, διότι έχουν σαφέστερους κανόνες για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε ένα θεμητό νόμιμο ανταγωνισμό, χωρίς τρευλώσεις και στρεφόμαστε ιδιαίτερα σε εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουμε υπόψη που δεν λειτουργούν <laughs> ιδιαίτερα καλά. Και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα για μια καλύτερη ενιαία εσωτερική αγορά με βελτιωμένους όρους. Ολοκληρώνοντα θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες της Γραμματείας θερμά. Συνολικά είχαμε τρεις ε, ε, συμβούλους, ε, ειδικού συμβούλους κατά τη διάρκεια της εργασίας και συνεργάστηκαν εξαιρετικά για την εκπόνηση της έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέγει ο Πρόεδρος και ευχαριστώ πολύ και η Μάσα. Πολύ σωστά. Λοιπόν, περνάμε αμέσως άμεσα στην ψηφοφορία. Τροπολογία 11. Όχοβα και Φόξ υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Και τροπολογία 10 του κυρίου Τριανταφυλλίδη υπέρ. Κατά απορρίφθηκε. Περνάμε στον συμβιβασμό 1 Όσοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Εγκρίθηκε. Και τώρα θα πάμε κατευθείαν στον συμβιβασμό 2. Υπέρ. Κατά. Εντάξει. Ας ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Συμβιβασμός 2. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για τον συμβιβασμό 2. Εγώ δεν θα συμμετάσχω στην ψηφοφορία. Εντάξει αλλάξατε άποψη. Εντάξει, τέλο πάντων. Ωραία. Λοιπόν, συμβιβασμός 2. Λοιπόν, εγείροντα τα σχήρα. υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 22 για διαγραφή. Διαγραφή από πλευρά Κορολά και Βόξ. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα εγκρίθηκε 20 ψήφοι υπέρ 13 εναντίον. Τροπολογία 23 τώρα, Κρόισμαν, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 24 αποσύρθηκε. Τροπολογία 25, Κουπάκης, Πουπάκης, υπέρ, της 25. Άρχεται η, τροπολο... η ψηφοφορία για την 25. Πέρας ψηφοφορίας ηλεκτρονικά για την 25 εγκρίθηκε 19 υπέρ 14 εναντίον. Συμβιβασμός 3 υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 29 με προφορική τροποποίηση που έχει τυπωθεί στον πίνακα ψηφοφορίας. Λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε αυτή την προφορική τροποποίηση. 29 με την προφορική τροποποίηση υπέρ κατά σαφώς εγκρίθηκε. Η τροπολογία 29 καταπίπτει χωρίς τροποποίηση και περνάμε στο συμβασμό 4 υπέρ κατά α, εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 35 του κυρίου Κρόιτσμαν Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Α, εγκρίθηκε. Ίντερ 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 5 υπέρ. Κατά. Και, αυτός, και αυτή η τροπολογία ε, εγκρίθηκε ο συμβιβασμός. Και περνάμε στην τροπολογία 39. Σωστό. Σωστό. Τροπολογία 39 του κυρίου Κρόισμαν υπέρ. Κατά απορρίφθηκε 40 κόρολα υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 41 Κρόιτσμαν υπέρ κατά ε, απορρίφθηκε αυτή της Βιομηχαν... Επιτροπής Βιομηχανίας αποκαλύπτεται 7 της Επιτροπής Βιομηχανίας ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίθηκε 42 για διαγραφή η τροπολογία 42. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε τη 42. Οι σοσιαλιστές έχουν έναν παραπάνω στην ψηφοφορία. Ας κλείσουμε όμως την ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε. Ένα α αποχωρήσει από την ομάδα του, των σοσιαλιστών που ψηφίζουν. Έχουμε και την ηλεκτρονική εποπτεία εδώ. Επόπτη ηλεκτρονικό εγκρίθηκε. 43, 44, 45 καταπίπτουν. Περνάμε στην 46. Υπέρ, παρακαλώ. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. 46 άρχεται η ψηφοφορία. The ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 20 υπέρ 14 ε, εναντίον. Ε, μία, μία ψήφος εναντίον 14 αποχές. Περνάμε στην επόμενη τροπολογία Κρόιτσμαν υπέρ κατά απορρίφθηκε. 47 στη συνέχεια. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τη 47. Έχουν έναν παραπάνω οι σοσιαλιστές πάλι να αφαιρεθεί ένα μέλος πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε 20 υπέρ 15 εναντίον τροπολογία 50 κόρολα τροπολογία 50 υπέρ θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε την 50 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε 20 ψήφοι υπέρ 15 εναντίον 49 ε, κρόσμαν καταπίπτει σύμφωνα με τις σημειώσεις μας και περνάμε και ψηφίζουμε την 51 Σάνδε Μόζε παρακαλώ υπέρ κατά εγκρίθηκε Επιτροπής Βιομηχανίας 5 υπέρ κατά εγκρίθηκε της Επιτροπής Παγκοσμίου Διεθνούς Εμπορίου 6 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 53, Σάντε υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Και περνάμε στην 52 προσθήκη, σωστό. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 52 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε 21 υπέρ 15 εναντίον. Τροπολογία 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 54 ηλεκτρονικά. 54. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 21 υπέρ, 15 εναντίον. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Περνάμε και πάμε στην τροπολογία 62 Σάντε Μόζε υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. 63 υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. 64 υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Ίντερ 1 υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Ίντερ 2, συγγνώμη. Ίντερ 2 εγκρίθηκε μάλιστα. Εντάξει. Ξέρατε για τι πράγμα έκανα λόγο και ψηφίσαμε. Είναι τα 4 καλύπτεται, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Είναι τα 5 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Είναι τα 10 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Είναι τα 7 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Και συμβιβασμός, ε, συγγνώμη, τροπολογία 65 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Περνάμε στην 26. 26α. Είναι η τροπολογία μου με προφορική τροποποίηση. Ο εισηγητής το κάνει δεκτό υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η 66 καταπίπτει, 67 του κυρίου Τριανταφυλλίδη υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 68 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Η 69 καταπίπτει, όχι είναι προσθήκη, 69 ως προσθήκη υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τη Επιτροπή Βιομηχανία η 11. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την Ήτρε 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Το ΕΛΚΑ έχει ένα μέλος παραπάνω τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και με τον έναν παραπάνω, έστω. Αλλά κάποιος να βγάλει την κάρτα του από το, το, μέλος παραπάνω. Τώρα, η επόμενη Κρόιτσμαν, υπέρ. Η 70 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Τροπολογία 71 κόρολα υπέρ κατά και αυτή εγκρίθηκε. Περνάμε στην 72 κόρολα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 72 τροπολογία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε 21 υπέρ 15 εναντίον. Η 13 καλύπτεται. Η 74 κόρολα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 74. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε με 22 υπέρ 14 κατά. Η 73 καταπίπτει. Συμβιβασμός 7 τώρα υπέρ κατά εγκρίθηκε. Της βιομηχανίας η 12. Επιτροπής βιομηχανίας 12 υπέρ Εντάξει, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 12. 12 Επιτροπής Βιομηχανίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε 21 υπέρ 14 εναντίον. Τροπολογία 77. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε αυτή. Και περνάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 3. Σάντε Μόζε υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Αιτιολογική σκέψη ε. Συμβιβασμό 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 9. Υπέρ. 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 9. Πέρας ψηφοφορίας Καταψηφίστηκε 14 υπέρ 23 εναντίον. Τροπολογία 1 για διαγραφή. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 1. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 22 υπέρ 15 εναντίον. Και περνάμε τώρα στο σχέδιο έκθεση στο σύνολό του που θα το ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση. Α, η τροπολογία 2. Α, είναι για την αιτιολογική σκέψη 15, τροπολογία 2 για διαγραφή. Άρχεται η ψηφοφορία για αυτή την αιτιολογική σκέψη. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 21-15. Έχουμε πάλι ένα μέλος του ΕΛΚ παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τώρα περνάμε στην ε, έκθεση γνωμοδότηση ως σύνολο. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Έχουν ένα παραπάνω μέλος το ΕΛΚ, από το ΕΛΚ. Κάποιος να βγάλει την κάρτα του από τη συσκευή. Εντάξει, καλύτερα τα πάμε τώρα. Τέλος ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα 36 υπέρ εγκρίθηκε λοιπόν και 2 εναντίον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σάντε Μόζε, πράγματι. None against Κανείς εναντίον, δύο αποχές, εντάξει, διορθώνει ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Προχωρούμε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 Προχωρούμε κυρίες και κύριοι σε αυτή τη σημαντική ψηφοφορία. Καταρχά θα ήθελα λίγη ησυχία για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε. Γιατί σας ε, λέω εξ αρχής ότι θα είναι δύσκολη και περίπλοκη η διαδικασία. Θα ζητήσω από τον εισηγητή κύριο Σβάμπε αν θέλει να πει κάτι στο ξεκίνημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό είναι που μου δίνετε το τον λόγο γιατί βεβαίως υπάρχει ενδιαφέρον εντό και εκτός Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, γραμματείας και της νομικής υπηρεσίας. Δεύτερον, μετά τις πολλές επικοδομητικές συναντήσεις με τους κοιοδησηγητές και μετά από πολλούς μήνες, καταλήξαμε στο ότι έχουμε ένα πακέτο από συμβαστικές λύσεις που αποτελείται από πέντε μέρη. Προσπάθησα λοιπόν να λάβω υπόψη ε, τις οποθετήσεις όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Εάν δείτε τις συμβαστικές προτάσεις ε, και το σχέδιο έκθεσης θα δείτε πως μετακινηθήκαμε σε πάρα πολλά σημεία και άρα αντικατοπτρίζει αυτό την άποψη της Επιτροπής Τρίτων. Ελπίζω λοιπόν και θέλω να το πω αυτό, πως το πακέτο αυτό άρα θα γίνει δεκτό από όλους ε, όσους ε, συνεισέφεραν ε, στη δημιουργία του. Η κοινή μας εργασία και οι κοινέ μας παραχωρήσεις θα πρέπει νομίζω να οδηγήσουν σε υιοθέτηση του πακέτου από όλους. Τεταρτόν μόνο στην δική μας επιτροπή θα κατευθύνταν πάνω από 1060 τροπολογίες. Έχετε τώρα 50 συμβαστικές ε, τροπολογίες ε, μπροστά σας και νομίζω πως ε, μπορούμε να ψηφίσουμε σε κάποιον ικανοποιητικό χρόνο και ελπίζω να μην χρειαστεί να ψηφίσουμε ακόμα σε 6,5 και να ακυρώσουμε την πίτσα που έχουμε παραγγείλει. Και μετά από συζήτηση πολλών ετών νομίζω καταλήγουμε σε ένα αποδεκτό αποτέλεσμα για να προωθήσουμε την εσωτερική αγορά προς συμφέρον των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ τον συγητή. Εάν συγκεντρωθούν όλοι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και θα ζητούσα από τον κύριο Σφάμπε και την κυρία Γκέπχαρτ να μου λένε νωρίς ε, είναι τι κατάσταση για να ξέρω αν θα πάμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία ή όχι. Αν εξ λοιπόν μου κάνετε νοήματα και δεν μιλάτε στα κινητά σας, θα προχωρήσουμε γρήγορα. Εντάξει κύριε Σβάμπερ. Λοιπόν, ξεκινούμε. Συμβιβαστική τροπολογία 2 για το άρθρο 1. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Για το άρθρο 1. Συμβιβαστική πρόταση για το άρθρο 1. Απλά η δική μου, ο δικός μου κατάλογος έλεγε 2. 398. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Άρθρο 2 σημείο 1. Συμβιβαστική τροπολογία για το 2-1. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Άρα προχωρούμε. 411. Τούρουνεν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ 23 κατά. δεν θα διαβάζω το, τις ψήφους εκτός αν κάποιος το θέλει. Επίσης μπορείτε να ψηφίζετε γρηγορότερα αν γίνεται. Πατά, πατάτε το κουμπί, τίποτα άλλο. Επόμενη συμβαστική τροπολογία. Άρθρο 2-2. 2-4. 2-2 διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ, κατά, δεκτή. Προχωρούμε. Συμβιβαστική τροπολογία η επόμενη. Για το άρθρο 2. 7. Συμβαστική 7. Υπέρ. Άρθρο 2 σημείο 3 υπέρ κατά δεκτή. Κύριε Τούρνεν, μήπως θα έλεγα να, να λέτε άρθρο και σημείο. Δεν έχουμε τους αριθμούς των συμβασικών τροπολογιών. Πείτε συμβαστική τροπολογία για το, άρθρο, για το άρθρο 2 παράγραφος 5 παραδείγματος χάρη. Σωστά, λέει ο πρόεδρος. Επόμενη συμβαστική τροπολογία άρθρο 2, σημείο 4 και αιτιολογική σκέψη 11α, 11β, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τώρα προχωρούμε. Συμβιβαστική τροπολογία για το άρθρο 2, σημείο 4, α, νέο. Παραπέρα. Πολύ καλή δουλειά κάνατε εδώ, κύριε Σιγητά. Άρθρο 2, 4, νέο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Προχωρούμε. Συμβαστική τροπολογία για το άρθρο 2, 5. Σημείο 5. Υπέρ. Κατά. Και αυτό είναι δεκτό. Συμβιβαστική τροπολογία για το άρθρο 2.5α νέο. Υπέρ. Κατά. Και αυτό είναι δεκτό. Προχωράμε με φοβερή ταχύτητα άρθρο 2, σημείο 6 και αιτιολογικές σκέψεις 12 και 13. Υπέρ, κατά και αυτό είναι δεκτό. Προχωρούμε. Τροπολογία 43 και Γιούρι 58. Υπέρ, κατά, δεκτή τροπολογία. Προχωρούμε. Τροπολογία 44 Διορθώνει ο πρόεδρος. Συμβιβαστική τροπολογία για το άρθρο 2 σημείο 8 και αιτιολογική σκέψη 14. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Προχωρούμε. Άρθρο, συμβαστική τροπολογία, άρθρο 2 σημείο 9 και αιτιολογική σκέψη 15. Δεν σας λέω σε ποια σελίδα είναι, γιατί ο καθένας έχει διαφορετική σελίδα. Στην 20. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προχωρούμε. Συμβαστική τροπολογία για το σημείο 11 και αιτιολογική σκέψη 16. 10 διορθώνει ο πρόεδρος και αιτιολογική σκέψη 16. Άρθρο 2 σημείο 10 και αιτιολογική σκέψη 16. πέρα. Άρθρο 2 σημείο 10 και αιτιολογική σκέψη 16. πέρα. Κατά δεκτή. Τροπολογία 60 της νομικής επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Προχωρούμε. Συμβιβαστική τροπολογία για το άρθρο 2 σημείο 11. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 46. μαζί με την Γιούρι 62. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Προχωρούμε. Η 491 καταπίπτει, τροπολογία 47 και η Γιούρι 63. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Προχωρούμε. 48 και Γιούρι 65. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική τροπολογία για το άρθρο 2 σημείο 16. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 66 της Νομικής Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική τροπολογία για το άρθρο 2.18. Σημείο 18. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Άρθρο 2 σημείο 19, τροπολογία 51 για διαγραφή. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική τροπολογία 2 σημείο 20. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Προχωρούμε. Τροπολογία 53. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία για την 53. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική τροπολογία για το άρθρο 3 και τα συναφή ε, κείμενα αιτιολογικών σκέψεων. Εδώ έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία από τους σοσιαλιστές. Θα ψηφίσουμε, θα πάρουμε όλο το κείμενο με, με την εξαίρεση των λέξεων χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα χρηματοοικονομικές υπηρεσίες άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Προχωρούμε. Καταπίπτουν όλες οι άλλες τροπολογίες για το άρθρο 3 που είναι πολλές σελίδες. Κύριε Τούρινεν, ξεχάσατε την 68 της νομικής επιτροπής. Και πού είναι αυτή, λέει ο πρόεδρος, στη σελίδα 27. Εμείς έχουμε την ίδια Η 68, σύμφωνα με τα δικά μου, ήταν κομμάτι της συμβαστικής τροπολογίας. Στο 2 σημείο 20. Εντάξει. Άρθρο 4. Εδώ υπάρχει συμβιβαστική τροπολογία για το άρθρο 4 και, τα, και τις συναφείς αιτιολογικές σκέψεις και έχει ζητηθεί ψηφοφορία σε έξι τμήματα. Συμβιβαστική τροπολογία 4 για το άρθρο 4 τμήμα 1 υπέρ. Κατά. 2 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτό το δεύτερο τμήμα. Τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Τέσσερα. Τέταρτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτό. Πέμπτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Έκτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Λάθος κουμπί πατήθηκε, τέλος πάντων, ξαναρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία και αυτό πέρασε. Προχωρούμε βασική τροπολογία το άρθρο 4α στη σελίδα 38 4α υπέρ κατά δεκτό. Φεύγουμε από το κεφάλαιο 1 λοιπόν. Ελπίζω να πάνε εξίσου γρήγορα και τα υπόλοιπα πρόεδρε. Εγώ έχω διάφορα πακετάκια εδώ. Έχουμε το κεφάλαιο 2 έτσι. Για συμβιβαστική 22 υπέρ κατά δεκτή. Οπότε περνάμε τώρα νομίζω. Πού πάμε. So we now go to compromise 20... Συμβαστική 23. Σελίδα 5. Συμβιβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε στην 673 την τροπολογία, σωστά. Πολύ καλή δουλειά εδώ κύριε Σίγητα. Um, Οπότε, νομίζω, ε, εκτός αν με διορθώσει ο εισηγητής, πάμε στα εκτιμώντας. Ε, μπορείτε να μου πείτε. Πάμε λοιπόν στα ανάλογα εκτιμώντας τώρα, σωστά. Οπότε περνάμε στα εκτιμώντας. Συμβιβαστική επί του 17. Συμφωνούμε όλοι. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 302 του κυρίου Μότη. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται και περνάμε στην 303 ροσφόρ πίπτη. Είμαστε στο άρθρο 6 άρα. Συμβιβαστική 24 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε στην 86 ροσφόρ. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Μετά. Τροπολογία 6, 9, 4, 5, 6 καταπίπτουν και η 100 της νομικών υποθέσεων. Μάλιστα. Οπότε περνάμε στην DR6 ή έχουμε τελειώσει. Ψηφίζουμε τίποτα άλλο. Are you sure? Είστε σίγουροι? Όχι. Τελειώσαμε με το δεύτερο κεφάλαιο. Γρήγορα πάμε. Περνάμε στο κεφάλαιο 3 λοιπόν. Συμβιβαστική 25. Παρακολουθείτε. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Οπότε περνάμε στο άρθρο 8. Καλά τα λέω. 88, 700 και τα λοιπά. Διαγραφή του άρθρου 8 υπέρ. Κατά. έχει δεκτή. Μετά περνάμε στην τροπολογία τη συμβιβαστική 26 υπέρ. Α, νομίζω θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Συμβαστική τροπολογία 26 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Οπότε περνάμε τώρα στην συνδυαστική επί του άρθρου 10. Εκτιμώντας 25 θέλετε να το ψηφίσουμε και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, Α, συγγνώμη, πρέπει να, πάμε πίσω, μου φαίνεται, να γυρίσουμε πίσω. Πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα την DR82. Ε, υπέρ. Κατά. Δεκτή. Και μετά πάμε και στην DR83. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 678 υπέρ. Κατά δεκτή. Και τώρα είμαστε στη συμβαστική τροπολογία επί της 25, το εκτιμώντας 25, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Οπότε είμαστε στην συμβαστική 27, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Οπότε περνάμε τώρα στην συμβαστική του άρθρου 11. Συμβιβαστική 28 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Περνάμε στην συμβιβαστική επί του άρθρου 12. χρειάζεται να ψηφίσουμε το εκτιμώντα 21 ή θεωρούμε πω υιοθετήθηκε με τη συμβιβαστική. Το αποτέλεσμα το ίδιο θα είναι, είμαι σίγουρο. Θέλετε να ψηφίσουμε. Όχι, το δέχεστε. Ωραία. Οπότε γίνεται δεκτό και το εκτιμώντα 21 και περνάμε στη συμβαστική 29 επί των άρθρων 11 και των εκτιμώντας 22 και 26 υπέρ. Κατά δεκτή. Περνάμε άρα στη συμβαστική τροπολογία επί του άρθρου 13. Σελίδα 23 στο δικό μου έγγραφο. Άρθρο 13. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Αυτή ήταν η συμβαστική τροπολογία 30. Και περνάμε στην 14. Επί του άρθρου 14. Η παριθμόν 31. Υπέρ. Κατά δεκτή. Οπότε πάμε στο σχέδιο στο DR106. Σωστά. Επί του άρθρου 15 υπέρ. Κατά δεκτή. Και μετά περνάμε στο 894 άρχεται η ψηφοφορία. και απορρίπτεται 13 υπέρ 24 εναντίον. Συμβαστική 32 επί το άρθρο 16 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Περνάμε αραστή τη συμβαστική επί το άρθρο 17 που είναι στη σελίδα 31. 32. Συμβιβαστική 33. 33. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 33. Α, έχουμε χωριστή ψηφοφορία, με συγχωρείτε. Άρχεται η ψηφοφορία στο πρώτο μέρος της συμβιβαστικής 33. Πέρας. Δεκτή. Μέρος δεύτερον. Τη συμβιβαστικής 33. Πέρας και αυτή δεκτή. Οπότε περνάμε στην DR114 επί του άρθρου 18 σελίδα 36 το δικό μου κείμενο DR114 υπέρ κατά δεκτή 115 υπέρ κατά τι. Συμβιβαστική 34 στο άρθρο 19 και τα σχετικά εκτιμώντας. Και πάλι τη ψηφοφορία ζητούν οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Δεκτή. Μέρος δεύτερο. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 22 έναντι 16. Οπότε περνάμε στην 140 της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του άρθρου 20. Άρθρο 20. Τζούρι 140 υπέρ κατά δεκτή σαφώς οπότε 126 με 128 κατά καταπίπτουν και πηγαίνουμε έχει διαγραφεί άρα το άρθρο 20 οπότε περνάμε στο 20α Οπότε, εκτός αν διαφωνεί ο εισηγητής, περνάμε στην 1053 για το νέο 20α. Συμφωνούμε, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1054, υπέρ, κατά, επίσης απορρίπτεται. Οπότε τελειώσαμε με άλλο ένα κεφάλαιο, καλά πάμε. Ε, we now move on. Τώρα περνάμε. Νομίζω στο κεφάλαιο 4, σωστό. Κεφάλαιο 4 μάλιστα. Λοιπόν. So all of this compromise on 21 falls. What about 105 now? 1057 η πρώτη που θα ψηφίσουμε υπέρ κατά απορρίφθηκε από ό,τι βλέπω επειδή υιοθετήθηκε η τροπολογία στο άρθρο 3 συμβαστική τροπολογία η συμβαστική και στο άρθρο 21 όλες οι άλλες καταπίπτουν και το 21 θα διαγραφεί επειδή καλύπτεται από το άρθρο 3. Σωστό, εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν όλες όσε σχετίζονται με το 21 οι τροπολογίες καταπίπτουν. Και περνάμε στο άρθρο 22 τώρα, σωστό. Άρθρο 22. Συμβιβαστική τροπολογία υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 1114. Σελίδα 13. Κυρία Ρόιτοβα. Υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα στον συμβιβασμό στο άρθρο 22α νέο. Όσοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίθηκε σαφές το αποτέλεσμα. Όλες οι άλλες τοπολογίες καταπίπτουν. Περνάμε στο συμβιβασμό στο άρθρο 23 υπέρ κατά εγκρίθηκε με κάθε σαφήνεια και περνάμε στην συμβιβαστική στο άρθρο 23α νέο στην σελίδα, την δική μου σελίδα στο κείμενό μου 17 συμβιβαστική στο 23α νέο άρχεται όσοι είναι υπέρ όσοι είναι υπέρ για το άρθρο αυτό κατά εγκρίθηκε σαφώς και περνάμε στο συμβιβασμό στο άρθρο 24. Υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Περνάμε στη συνέχεια στην 1176. Είναι αρκετά πιο κάτω. Στην σελίδα 26 στο κείμενό μου. 1176 και 1178 ταυτόσημες ψηφίζουμε υπέρ αυτών κατά απορρίφθηκαν αυτές οι δύο Βάις δεν θα ψηφιστεί όχι η ίδια περίπτωση Συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσουμε την 1178, σφάλμα μου, ζητώ συγγνώμη, 1178 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε σαφώς. 1177-1179 δεν θα ψηφιστούν. ...1180 δεν θα την ψηφίσουμε. Τι λέτε εσείς. All Λοιπόν, θα ψηφίσουμε την 1180 για να είμαστε σίγουροι υπέρ κατά. Απορρίφθηκε σαφώς. 358 Ροσφόρ υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 358. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Και η 146 του κ. Σβάμπ υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Σαλβίνη, Σαλβίνη, τροπολογία ως προσθήκη, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 23 του κ. Σουβάμπ, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τρεις ταυτόσημες, η 1406, 1411 και η 1412, η... άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε αυτές τις τρεις τροπολογίες. Πέρας ψηφοφορίας, Αποτέλεσμα απορρίφθηκαν και οι τρεις απορρίφθηκαν αυτές οι τρεις. Η 1406 το Α, καταπίπτει, εντάξει. Καταπίπτει. It says that because you can't have an addition because you've. No, it's rejected. Mm -hmm you rejected this, so you can't have an addition to it. Okay, you can have an alternative. You can have an alternative, right. So 118. Λοιπόν, η επόμενη είναι 1182, εντάξει. Ψηφίζουμε λοιπόν. 1182, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε λοιπόν. Η 362, Σαλβίνη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Η 363 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε λοιπόν. 19-19 ισοψηφία, μία αποχή. ισοψηφία απορρίπτεται. Η Συμβαστική τροπολογία στο 26, σε τμήματα η ψηφοφορία που ζητήθηκε από την Ενωτική Αριστερά και τη Βόρεια Πράσινη Αριστερά. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, και αυτό εγκρίθηκε. Και έτσι οι τροπολογία στο άρθρο 26, οι υπόλοιπε καταπίπτουν. Και περνάμε αμέσως στο 27. Σελίδα 45 παρακαλώ. Μάλιστα. Διασπάθηση χάρτου. Λοιπόν, σελίδα 44 σε σχέση με το κείμενο μου. Συμβαστική τροπολογία στο 27. Όσοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Και τώρα περνάμε κατευθείαν στο άρθρο 28. Συμβαστική τροπολογία. Το δικό μου κείμενο στη σελίδα 47. Συμβαστική στο άρθρο 28. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Σαφώς. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία. 1378. Όλες οι άλλες τροπολογίες του 28 καταπίπτουν. Ψηφίζουμε την 1178 Weisgerber υπέρ κατά εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο συμβιβασμό στο άρθρο 29 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 1441 Α, ολοκληρώσαμε λέτε, καταπίπτει αυτή. Από ό,τι φαίνεται ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο 4. Chapter 5, we have no votes on Exactly, yeah. But just note that the jury members are deemed adopted pursuant to Rule 15. Uh, so, uh, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για τα πρακτικά, το κεφάλαιο 5 Ενισχυμένη συνεργασία με την ε, νομική επιτροπή γίνεται δεκτή χωρίς να ψηφίσουμε. Όλο το κεφάλαιο 5 εγκρίνεται με τη διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας. Τελευταίο κεφάλαιο, έτσι. Κεφάλαιο 6. Α, υπάρχει και το 7. Άλλα δύο κεφάλαια. Άρθρο 40 τέσσερι τροπολογίε για διαγραφή. Για διαγραφή υπέρ, κατά, αποχέ, φεύγει το 40. Άρα και τα συναφή, και οι συναφείς αιτιολογικέ σκέψει σε εξορισμό, αν δεν ψηφίσουμε. Άρθρο 41. 151, 15-18 Γκέπχαρντ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 15-19. Γκέπχαλτ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 19-19. Ένα άτομο δεν ψήφισε. Λίγο πιο γρήγορα. Μια σειρά του απολογιών Κάρας. 15-20, 15-21, 22-23. Ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 15-24. Κοράτσα Μπίλ και Καλνιέτε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 18 προς 20. Έχει αποσυρθεί η 1525 του κ. Κρόιτσμαν. Συμβιβαστική για τη 45α για το 44 υπέρ κατά δεκτό. συμβιβαστική 45 46 τώρα υπέρ κατά δεκτή. 173 για το άρθρο 46. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβαστική 48. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Και τι αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη εγκρίνεται. 49 συμβαστική υπέρ. Κατά. Δεκτή. εγκρίνεται η 33 389 Ιβάνοβα για τι θετολογική σκέψη υπέρ κατά δεκτή εκόν 9 άρχιρη ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 18 προς 15 η 8 της Οικονομικής Επιτροπής Τέλο πάντων, ε, με τα χέρια. Ποιοι είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Ωραία. Κεφάλαιο 7. «191 της νομικής επιτροπής» κατά δεκτή. Η 49 συμβαστική εγκρίθηκε, αλλά δεν ψηφίζουμε για την 34. Άρθρο 48. Μέντες. Υποβλήθηκε χτες ε, προφορική τροπολογία για τη 49 η προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας Πέραση Δεκτή. Τρία Τούρνεν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 396. Ράπτη Πουπάκης. Άρχεται η ψηφοφορία για την 396. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 50. Στο παράδειγμα 1 τμήμα α. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Άρα όλα τα τμήματα του παρήματος 1 τμήμα α 51 συμβαστική για το τμήμα Β υπέρ, κατά, δεκτή. Τα υπόλοιπα καλύπτονται από την ε, το συμβαστική αυτή, έτσι δεν είναι. Όλες οι επόμενες καλύπτονται από το, τη συμβαστική αυτή. Αιτιολογική σκέψη 2. 216 τροπολογία νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε τώρα. 216, 217 και έκον 1. Για να τα... Υπάρχει συμβιβαστική 1 για την αιτιολογική σκέψη 2. Δεν το έχουμε. Αλλά πρέπει, έπρεπε να το έχουμε. Σωστά. Λοιπόν, συμβιβαστική 1 για την αιτιολογική σκέψη 2. Ψηφίζουμε. Που καλύπτει την αιτιολογική σκέψη 2. Συμφωνείτε. Έχει γίνει λάθος, λέει ο, ο πρόεδρος. Θέλω να το ξεκαθαρίσω με τον εισηγητή και του σκιώδης. Εγώ έχω καταλάβει το εξή. Στις αιτιολογικές σκέψεις όταν τελειώσει το παράδειγμα 3, παράγραφος 4, 4 δέλτα. Πάμε από το παράδειγμα 3 στις αιτιολογικές σκέψεις. Εγώ δεν έχω σελίδες. Οι 2.16, 2.17, 2.15 και έκον 1. Με καταλαβαίνετε που, που είμαι. Υπάρχει μια συμβαστική πρόταση που δεν έχετε μπροστά σα για την αιτιολογική σκέψη 2 που καλύπτει και τι τέσσερι τροπολογίε και, και έχει συμφωνηθεί με τον εισηγητή. Ψηφίζουμε λοιπόν την, την, την ε, συμβαστική για, το για την αιτιολογική σκέψη 2. Υπέρ, κατά, δεκτή. Αιτιολογική σκέψη 3. Τέσσερα. 220, 221 Τούρνεν. Για τη 221 ψηφίζουμε πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 225 και 226 ίδιες. Τούρνεν και Ροσφόρ αντίστοιχα. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για αυτές τις δύο τροπολογίες. Πέρας ψηφοφορίας δεκτές 227 ήταν γλωσσική δεν ψηφίζεται 228 Τούρνεν. άρχεται η ψηφοφορία για την 228 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 18-21 229 να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για τη 229 καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Ψηφίζουμε το κείμενο συνολικά. Σωστά κύριε Σιγητά, κύριε Γκέπχαρτ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σβάμπ για την πολλή δουλειά που έχει κάνει. Την κάναμε όλοι από κοινού, γιατί πραγματικά δεν ήταν τίποτα το εύκολο αυτό που κάναμε. καθώς ε, το κείμενο της Κομισιόν ήταν προβληματικό και θα ήθελα μετά να παρατηρήσω πως στο μέλλον θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτούς και βλέπω πως συγκατανεύει ο κύριος Σβάμπ Όσο όταν έχουμε τόσο άσχημες προτάσεις στο μέλλον, δεν θα αποδεχόμαστε καν να εργαστούμε από αυτόν. Και θα αναπέμπουμε το κείμενο κατευθείαν. Αυτό ήθελα να πω. Δεύτερον, και λυπούμε γι' αυτό γιατί πέρασα πάρα πολλές ώρες, πάρα πολλή δουλειά για το ότι πρέπει να συστήσω στην ομάδα μου μετά τη χτεσινή συζήτηση να καταψηφίσουμε αυτόν τον συμβιβασμό. Θα είμαστε κατά στην ψηφοφορία και θα ήθελα να αιτιολογήσω γιατί συνέβη αυτό, γιατί ε, μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου αυτή την εντολή χτες για να το ξέρουν και οι άλλες ομάδες. Είχε πει ευθύ εξ αρχή η ομάδα μου πως δεν μπορούμε να δεχτούμε κανένα κείμενο στο οποίο και μία ακόμη πρόταση θα σήμαινε επιδείνωση της προστασίας των καλλιτών σε ένα έστω κράτος Και αυτό εδώ πέρα έχει συμβεί. Μπορώ να σας αναφέρω 5-6 παραδείγματα έτσι πρόχειρα. Αλλά τόσο αν δεν θέλω να μακρηγορήσω θα περιοριστώ σε δύο μόνο. Για να εξηγήσω γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε πρώτα απ' όλα και αυτό το είχαμε πει ευθύς εξ αρχής, είναι πως η ομάδα, μας, η ομάδα μας δεν μπορεί να αποδεκτεί πως η υπηρεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ολόκληρη έχει φύγει εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Βγάλαμε κάποια κομμάτια και συμφωνήσαμε καθώς είχαν καλυφθεί αυτά σε άλλες οδηγίες, π.χ. μέσω της οδηγίας δικαιωμάτων των καταναλωτών, αλλά... Ε, καταναλωτικής πίστης, με συγχωρείτε. Αλλά υπάρχουν κομμάτια τα οποία δεν ε, καλύπτονται και εδώ πέρα μιλάμε για τη μικρή καταναλωτική πίστη και εδώ πέρα βεβαίως υπάρχει ο συνάδελφος ο οποίος μας είπε πως ε, κύριος πως στην Σκανδιναβία υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τις πολύ μικρές συμβάσεις δανειακές μέσω SMS οι οποίες δεν καλύπτονται από την οδηγία και επειδή βγάλαμε τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν καλύπτονται ούτε από την οδηγία δικαιωμάτων των καταναλωτών. Οπότε το δικαίωμα υπαναχώρησης και άλλα τα οποία εμείς ως σοσιαλδημοκράτες θέλαμε εδώ πέρα δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εγγύησης και αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα για την ομάδα μου. Ένα δεύτερο πρόβλημα και κυρίως επειδή στον τομέα αυτών προβλέπεται μια πλήρης εναρμόνιση, δηλαδή δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο τα κράτη-μέλη περαιτέρω στον τομέα αυτών, γιατί μιλάμε για πλήρη εναρμόνιση. Αν είχαμε ελάχιστη εναρμόνιση θα ήταν καλό και αυτό ζητούσαμε βεβαίως πάντα και θα το είχαμε δεχτεί. Ένα δεύτερο παράδειγμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και το λέω εδώ και εβδομάδες είναι πως το άρθρο 10 η ομάδα μου δεν μπορεί να αποδεχτεί πλήρη εναρμόνιση γιατί η διατύπωση που έχετε εκεί πέρα δεν είναι αποδεκτή απλά από την ομάδα μου γιατί το θέμα εδώ πέρα είναι το ότι όταν μιλάμε για συμβάσεις εκτός της ε, οικίας ε, μπορούν ε, να γίνουν αυτές με γραπτή μορφή μόνο μετά από αίτημα του καταναλωτή και μάλιστα αναφέρεται σε αυτό το άρθρο πως ο καταναλωτής θα πρέπει να ζητήσει την σύμβαση για να τη λάβει και μιλάμε μετά για διαρκές μέσο αποθήκευσης δηλαδή δεν μιλάμε καν για χαρτί μπορεί να είναι σε ένα USB ή ένα CD-ROM κάτι το οποίο βεβαίω δεν μπορεί να το εξετάσει ούτως ή άλλως ε, κάποιος ε, στα ορθιά το τι ακριβώς του είπε ο πολιτής. Και ακριβώς εκεί πέρα έχουμε αυτή τη διατύπωση στα αγγλικά θα δοθεί στον καταναλωτή σε διαρκές μέσο στο μέτρο που αυτό θεωρείται κατάλληλο δεδομένης της φύσης του, της σύμβασης. Όχι, δεν είναι αποδεκτό αυτό. Εδώ πέρα ανοίγει διάπλατα η πόρτα για να πει κάποιος «Α, εμείς ε, δεν χρειαζόμαστε σε αυτή την περίπτωση γραπτή σύμβαση». Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν δέχεται η ομάδα μας. Είναι κάτι το διασφαλισμένο σε πολλά κράτη-μέλη μέσω κανόνων ε, του εθνικού δικαίου που θα πρέπει να καταργηθούν γιατί στον τομέα αυτών επίσης προβλέπεται πλήρης εναρμόνιση. Αυτά είναι δύο παραδείγματα τα οποία μας ε, οδηγούν στο να μην ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ωραία. Πρέπει να περάσουμε στην τελική ψηφοφορία, αλλά δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσει τίποτα σύγκριτης. Όχι. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Επί της πρότασης της Κομισιόν, όπως αυτή τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιοι δεν θέλουν να ψηφίσουν, βλέπω. 38 ψηφίζουν αυτή τη στιγμή. Να, κάποιοι ακόμα. Οπότε γίνεται δεκτή. 22 υπέρ, 16 κατά μία αποχή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νομίζω πως ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν είχαμε ε, πλήρη πλειοψηφία από πλευράς ε, εισηγητή. Νομίζω πως ε, το κείμενο πολύπλοκο και θα χρειαστεί βεβαίως προσοχή πριν πάει στην Ολομέλεια. Ψηφίσαμε ήδη την πρόταση. Ξέρω πως θέλει να τα κάνει όλα αυτά ο εισηγητής, αλλά θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί χωρίς τη δουλειά αυτή για να καταλήξουμε συμβαστικές προτάσεις θα είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ψηφοφορία. Πράγματι έχει δίκιο η κυρία Γκέπχαρτο να λέει πως στο μέλλον ε, δεν πρέπει να τα δεχόμαστε έτσι αυτά τα κείμενα. Βεβαίως θα μπορούσαμε να πούμε πως και η Κομισιόν θα μπορούσε να είναι πιο επικριτική για το έργο της προηγούμενης Επιτροπής. Σε πάση περιπτώσει τώρα έχουμε κάτι θα αποτελέσει βάση για να δουλέψουμε και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και Λοιπόν, τελειώσαμε άρα με την συνεδρίαση. Να πω όμως πώς ε, προτείνουμε στους ηγητές και σκιώδες να χρησιμοποιήσετε αυτή την αίθουσα με διερμηνία για τα υπόλοιπα 35 λεπτά για συνέντευξη τύπου εάν θέλετε κάτι τέτοιο γιατί αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει ενδιαφέρον και η υπηρεσία τύπου έχει οργανώσει συνέντευξη τύπου. Όσοι λοιπόν θέλουν να λάβουν μέρος μπορούν να μείνουν, να ανέβουν εδώ πέρα στο βήμα. Η διερμηνία υπάρχει. Οπότε θα ζητήσω από τους υπόλοιπους συναδέλφους να φύγουν. Να πω πως συνεδριάζουμε την ερχόμενη εβδομάδα 3 η ώρα. Στις 10 ε, του μηνός. Ευχαριστώ.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 Uh, Οπότε κυρίε και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη τύπου. Να προσκαλέσω και τους και ηγητές που θέλουν να έρθουν στο βήμα. Κυρία Γκέπχαρτ είναι εδώ. Α, είναι έξω. Θα έρθει. Κυρία Τούρινεν, Έμιλι. I think so. Mr. Rochefort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 Uh, uh, Καλησπέρα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όσους είναι στην αίθουσα και σε όσους παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Νομίζω μεταδίδονται και στην αίθουσα τύπου αυτά. Οπότε, για όσους δεν είδαν τη μετάδοση, είμαι ο Μάλκομ Χάρμπορ, πρόεδρος της Επιτροπής Ιστορικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να δώσουμε μια πρώτη αντίδραση για την ψηφοφορία για την οδηγία δικαιωμάτων καταναλωτών που προηγήθηκε. Οπότε ο εισηγητής, ε, ο Αντριος και ο εισηγητές, ε, ε, κυρία... Οι εκπρόσωποι των σοσιαλιστών, φιλελευθέρων και πρασίνων και μετά βέβαια θα δεχτούμε ερωτήσεις ε, από τους παρόντες. Υπάρχει κάποιος? Ωραία. Απλά λοιπόν πρόκειται για μια ενημέρωση. Οπότε θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να υπενθυμίσω στους ε, θέατες μας πως μπορείτε να λάβετε το ενημερωτικό μας δελτίο. Βρίσκεται στο διαδίκτυο και βλέπετε και ένα δίκτυο τους φίλους της ΙΜΚΟ και μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε τακτικά νέα. Οπότε θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή για να μας πει την άποψη έχει τη η πλειοψηφία, ψηφοφορία και ε, ποια είναι τα επόμενα βήματα για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Ε, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχήν με ανακουφίζει ιδιαίτερα πάρα πολλοί από τους συμβιβασμούς που ψηφίστηκαν σήμερα υπερκομματικά εγκρίθηκαν και έτσι έχουμε ευρεία συνένεση, μας υποστηρίζουν ευρέως στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Μπορούμε να το πούμε μετά από αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτή την μεγάλη υποστήριξη θα έχουμε. Φυσικά θλίβομαι ιδιαίτερα ότι στο τέλος στην ψηφοφορία δεν είχαμε τόσο μεγάλη πλειοψηφία. Όμως αυτό συμβαίνει στην πολιτική ζωή καμιά φορά να πρέπει να λαμβάνεται μία απόφαση και υπό αυτού του όρου. Και έτσι σέβομαι το ότι άλλε κοινοβουλευτικέ ομάδε δεν μπόρεσαν αυτό το συμβιβασμό να τον υπερψηφίσουν στο τέλο. Θλίβομαι γι' αυτό, αλλά το δέχομαι το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ο συμβιβασμό που πλειοψηφικά εγκρίναμε και η πλειοψηφία ήταν επαρκώ σαφή, δύο σημαντικέ βελτιώσει συνεπάγεται για την ε, ευρωπαϊκή αγορά. Η ψηφιακή εσωτερική αγορά, η αγορά μέσω homepages και online διαδικτυακά, τα τελευταία έξι χρόνια διπλασιάστηκε. Αυτό είναι μια σημαντική συνεισφορά μακροπρόθεσμα για την εξέλιξη της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Καταναλωτές όλο και περισσότερο νέοι, όλο και περισσότερο διασυνοριακά αγοράζουν και ακριβώς νέοι που όχι μόνο σε ένα σημείο αλλά και στο εξωτερικό καταρτίζονται, εκπαιδεύονται, φοιτούν και υστερότερα στη συνέχεια εργάζονται. Για αυτούς είναι πολύ σημαντικό σε μια ενιαία εσωτερική αγορά να έχουμε ενιαίου κανόνες για αυτή την αγορά. Ιδιαίτερα πιστεύω ότι το δικαίωμα ανάκληση που το έχουμε εναρμονίσει όσον αφορά τη διάρκεια του με όλες τις εξαιρέσεις και με όλες τις άλλες προϋποθέσεις και όρους που θα ισχύουν σημαντικά συνεισφέρει την ενίσχυση αυτής της διασυνοριακής δυνατότητας εμπορίου στο διαδίκτυο online, ηλεκτρονικά. Σημαντικό είναι να έχουμε και την προστασία καταναλωτών που την αναλύσαμε σε όλες τις συνιστώσεις σχετικά και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν υπάρχει επιδείνωση του δικαίου του δικαιώματος προστασίας καταναλωτών σε κανένα σημείο. Ίσως σε επικάλυψη με άλλες οδηγίες μπορούν να υπάρχουν ερωτήματα που στη συνέχεια μπορούν να αποσαφινιστούν. Ε, προηγούμενα αναφέρθηκε ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν μικροπιστώσεις ή δάνεια που δεν καλύπτονται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα του ελάχιστου εναρμονισμού της οδηγίας υπαροχής υπηρεσιών για τους καταναλωτές. Εδώ πιστεύω ότι κατεπηγόντως πρέπει για τους καταναλωτές να ληφθούν μέτρα πανευρωπαϊκά, ώστε έτσι δεν θα υπάρχει κάποια διαφωνία επ' αυτού. Και δεύτερον, συμβαίνει το εξή με αυτή την οδηγία. Σε καμιά φορά η πορεία, η οδός για την προστασία καταναλωτών αφενός και αφετέρου η δυνατότητα να έχουν οι καταναλωτές παροχή υπηρεσιών χωρίς προσκόμματα και εμπόδια έπρεπε να ισορροπηθούν, να εξισορροπηθούν. Είναι μια απόφαση που δεν ήταν εύκολο, καθόλου εύκολο να ληφθεί. Βρήκαμε όμως νομίζω τη σωστή πορεία για να το κάνουμε αυτό. Συνοψίζω, προστασία καταναλωτού στο ανώτατο επίπεδο και ελευθερίες για την εσωτερική αγορά που συμβαδίζουν. Γι' αυτό με ανακουφίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορία. και ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουμε καλή συνέχεια και πρόοδο για αυτά τα θέματα με αυτές τις ρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Uh, um, Ευχαριστούμε. Οι σκιώδεις εισηγητές, καταρχάς η κυρία Γκέπχαρτ. Η κυρία Κέφαντε, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και εγώ ίδια αισθάνομαι ανακούφιση διότι ελήφθη αυτή η απόφαση με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και αν δεν μπόρεσα να υπερψηφίσω αυτή την απόφαση. Διότι <clears throat> Πρέπει αφενός να πω ότι είχαμε μια πολύ προβληματική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιτραπέζης που εξετάζαμε και το κυριότερο πρόβλημα είναι μέσω αυτής της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τα κράτη-μέλη <clears throat> δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν θα έχουν τη δυνατότητα αυτή το τελώς να ρυθμίζουν κάποιους τομείς όπου θα ήταν αναγκαίο να προβούν τα κράτη σε δικές τους ρυθμίσεις εκεί όπου θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να το κάνουν. Νομίζω σε αυτόν τον τομέα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Η δική μου ομάδα, η σοσιαλδημοκρατική ομάδα, όπως είχε αυτή η πρόταση τραπέζης... δεν μπόρεσε να την υπερψηφίσει. Και αυτό επειδή σε διάφορους τομείς λιγότερα δικαιώματα απορρέουν στο τέλος τέλος ω τελικό, τελικό αποτέλεσμα από ότι αυτά τα οποία διασφαλίζονται σήμερα στα κράτη-μέλη. Ένα από τα παραδείγματα είναι πράγματι ο τομέα τη παροχή οικονομικών υπηρεσιών, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που δυστυχώ συνολικά έχει εξαιρεθεί από την οδηγία περί παροχή υπηρεσιών. Αυτό δεν μπόρεσα να το δεχτώ. Μέχρι τελευταίου λεπτού αγωνίστηκα να προσπαθήσω να πείσω τον κύριο Σουβάμ για το γεγονό ότι δεν θα έπρεπε να εξαιρεθούν αυτέ οι υπηρεσίε από το πλαίσιο αυτό. Δεν το κατάφερα όμω να το πετύχω. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η χορήγηση πιστώσεων όσον αφορά την ε, οδηγία περί πιστώσεων προς τους καταναλωτές, συγγνώμη γιατί είναι δύσκολη η ορολογία για αυτό τον, του τίτλου αυτού, θα αρχίσει να ισχύει από ένα συγκεκριμένο επίπεδο συγκεκριμένα και χειροπιαστά. Για ένα επίπεδο κάτω από αυτό, επειδή σε αυτόν τον τομέα είχαμε ελάχιστε ενερμονήσει, ε, εντασσόμεθα στι ε, τομεακέ οδηγίε που τώρα θα αντικατασταθούν από αυτή την οδηγία που θα έχουμε στη διάθεσή μα. Αυτό σημαίνει ότι εκείνοι που δεν θα βρίσκονται σε αυτή την οδηγία για τις πιστώσεις καταναλωτών και που δεν θα καλύπτονται από τα δικαιώματα καταναλωτών, όλα τα δικαιώματα καταναλωτών που θα είχαν, ιδίω το, δικαίωμα ανάκλησης, δεν θα ενταχθούν. Και δεν είναι σαφές τι θα γίνει με αυτά τα δικαιώματα. Πρόκειται κατά κανόνα για πολύ μικρές ε, πιστώσεις, 20, 30, 50 ευρώ ως ποσά που προσφέρονται στους νέους εφόσον είναι νεότεροι από 18 έτη τότε ισχύει η νομοθεσία περί ανηλίκων. Αν όμως είναι πάνω από 18 και έχουν αρκετά τέτοια ε, ποσά ως πιστώσεις μπορούν να έχουν προβλήματα. Δεν θα έχουν δικαίωμα ανάκλησης, δεν θα έχουν σαφή πληροφόρηση τι θα συμβαίνει όσον αφορά το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο κτλ. Αυτά είναι προβληματικά θέματα και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μπόρεσα να δεχτώ και να υπερψηφίσω την πρόταση. Δεν μπόρεσα επίση να δεχτώ και κάτι άλλο. Στου τομεί εκείνου όπου πρόκειται για πληροφορίε που θα πρέπει να διατίθενται, δηλαδή άρθρα 10 και 11, ένα πλήρη εναρμονισμό προβλέπεται. Ενώ βλέπουμε ότι έχουμε πολύ γενικόλογε διατυπώσει ε, σε σχέση με αυτά τα άρθρα. Αφενό με προβλέπεται βέβαια ότι οι επιχειρήσει όταν θα έχουν ε, τέτοιου είδους συναλλαγές ε, στο κατόφλι κάποιου νοικοκυριού Τώρα ε, ε, δουλεύουμε στα αγγλικά και δεν θυμάμαι σωστά τη γερμανική ορολογία. Αν δεν είναι εύθετο για το, μια τέτοια σύμβαση, μπορεί να υπάρξει ε, η παρέκκληση από τη σύναψη γραπτών συμβάσεων. Αυτό το βρίσκω πολύ προβληματικό. Πολύ προβληματικό, διότι όταν έρχεται η ώρα και η στιγμή σε κάποια κράτη-μέλη να γίνεται αυτό, αυτόματα τότε συμβαίνει ότι μια τέτοια σύμβαση πρέπει γραπτό να είναι δεδομένη με υπογραφή κιόλα, ώστε να ισχύει το συμβόλαιο, η σύμβαση Γιατί Τώρα στο κείμενο κείμενο το οποίο ψηφίστηκε και εγκρίθηκε, αυτό παίρνει σχετική αξία. Έχει ο έμπορο την δυνατότητα να πει Α, είναι έκτακτη αυτή η περίπτωση και γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε γραπτέ συμβάσει. Γνωρίζει αυτή Δεν γνωρίζει όμω ο καταναλωτή αυτή την έκτακτη ειδική κατάσταση και δεν ξέρει πώ να την αντιμετωπίσει. Δεν ξέρει κατά κανόν όμω θα είχε δικαίωμα να ζητήσει μια γραπτή σύμβαση και ότι μπορεί να απαιτήσει να υπάρξει γραπτή διατύπωση. Αυτά όλα είναι στοιχεία που αποδεικνύουν γιατί η ομάδα μου ψήφισε όπω ψήφισε. Για γιατί δεν δεχτήκαμε αυτό το οποίο προτάθηκε. Θα μπορούσαμε ενδεχόμενα να το είχαμε δεχτεί αν σε αυτόν τον τομέα ένα ελάχιστο εναρμονισμό είχε προβλεφθεί ω δυνατότητα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν το περαιτέρω δίκαιο το οποίο θα μπορούσε να καλύπτει τέτοιε περιπτώσει να το διασφαλίζουν από πλευρά του. Αυτό όμω δεν προβλεπόταν από αυτή τη συμφωνία και γι' αυτό αυτό ήταν κάτι απόλυτα απαράδεκτο. Τώρα, ωστόσο, από την άλλη πλευρά, με ιδιαίτερη ε, ευχαρίστηση άκουσα, με πληροφόρησαν ότι προφανώ ο κύριο εισηγητή ακριβώ υπέβαλε την πρόταση μέχρι την Ολομέλεια να ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα. Μα προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Και ίσω να υπάρξουν και κάποιε δυνατότητε βελτιώσεων μέχρι τότε. Φυσικά είμαι πρόθυμη να κάνω χρήση αυτή τη προσφορά. Και αν καταφέρουμε στο τέλο τέλο να έχουμε κάποιε καλέ, καλύτερε διατάξει που θα ε, διαπραγματευτούμε μέχρι την Ολομέλεια, τότε φυσικά δεν θα ε, σταματήσω την πορεία των πραγμάτων, δεν θα είμαι εναντίον, διότι υπάρχει εδώ κάθε θεμητό δικαίωμα έναντι των καταναλωτών να υπάρξει αυτή η προστασία. Αυτό που θέλω είναι με την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών να έχουμε πρόσθετη αξία υπέρ της προστασίας των καταναλωτών και να μας εμπνέει και να μας διέπει η φιλοσοφική αρχή ότι όταν κάνουμε λόγο για τέτοια δικαιώματα καταναλωτών θα πρόκειται κυριολεκτικά για δικαιώματα καταναλωτών και όχι πρώτα και κύρια για την ενιαία εσωτερική αγορά όπως αποκόμισα την εντύπωση από πρώτο χέρι συζητήσεις. Δηλαδή η πόρτα είναι ανοιχτή, η πύλη είναι ανοιχτή για περαιτέρω βελτιώσει μέχρι την Ολομέλεια. Προσδοκώ και προσβλέπω να δω τι θα γίνει, τι θα καταφέρουμε να πετύχουμε σε αυτόν τον τομέα. Όχι μόνο σε αυτού του δύο τομεί που προανέφερα, αλλά και στου άλλου τομεί που απομένουν και στου οποίου εμεί θέλουμε, δεν μπορέσαμε να δεχτούμε του συμβιβασμού, επειδή δεν ήταν μόνο δύο από του συμβιβασμού, αλλά πέντε ε, του οποίου δεν μπορούσαμε να δεχθούμε, επειδή παρόμοια προβλήματα ετίθεντο για μα. Αλλά δεν θέλω να μονοπολίσω το χρόνο, ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ, ε, ο κύριο Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, σήμερα το πρωί ξαναδιάβασα το αρχικό κείμενο της ε, πρότασης ε, οδηγίας της Επιτροπής, κείμενο του Οκτωβρίου του 2008. Πήγαμε, περάσαμε πολύ μακρύ δρόμο έκτοτε. Το κείμενο αυτό ήταν ένα κακό κείμενο, όντως κακό, που έβλεπε τα θέματα του καταναλωτή με μια ελαφρότητα που έρχονταν σε αντίθεση με το σύνθετο χαρακτήρα της κατανάλωσης σήμερα στην κοινωνία μας, αλλά και το ουσιαστικό και το ότι έγινε ουσιαστικό στοιχείο της οικονομίας και της ζωής των Ευρωπαίων αλλά και της καθημερινότητας της Ευρώπης, ανεξάρτητα από τη χώρα, το επίπεδο ζωής ή την ηλικία του. Η κατανάλωση είναι βασικό χαρακτηριστικό της καθημερινής ζωής. Η οδηγία αυτή δεν είναι τέλεια. Ακόμα και μετά την ψηφοφορία που είχαμε, το σχέδιο οδηγία δεν είναι τέλειο. Λαμβάνοντα υπόψη το από πού ξεκινήσαμε. Θέλω ωστόσο πραγματικά να αποτίσω φόρο τιμή στον ε, κύριο Σφάμπε, τον εισηγητή, διότι έκανε ε, αλλά και στις ομάδες που τον υποστήριξαν και τις τεχνικές ομάδες της Επιτροπής, αλλά και εμάς, τους σκιώδεις εισηγητές, επιτρέψτε μου να πούμε. Δουλέψαμε πολύ για να βελτιώσουμε το κείμενο και θα ήθελα να σας ζητήσω να συγκρίνετε το αρχικό κείμενο με αυτό που ψηφίστηκε σήμερα στην Επιτροπή. Θέλω να πω ότι η οδηγία αυτή προασπίζει τους καταναλωτές. Να δηλώσω επίσης ότι βελτιώνει την ικανοποίηση των καταναλωτών του καταναλωτή και των δικαιωμάτων περιλαμβάνει δύο πράγματα. Και τα δικαιώματα, αλλά και την καλύτερη αγορά, την, την αγορά με καλύτερη τιμή και την βέλτιστη ποιότητα. Πολλοί το ανέφεραν. Ένα νέο φαινόμενο που ζούμε σήμερα, που εμφανίζεται με ηλικιώδη ταχύτητα, είναι η δυνατότητα αγοράς στο ίντερνετ καταναλωτικών προϊόντων. Εδώ δεν υπάρχουν σύνορα. Αυτό ταυτόχρονα μας μαγεύει τους Ευρωπαίους να ανοίγουμε την αγορά μας αλλά και μας τρομοκρατεί ταυτόχρονα διότι υπάρχουν τόσα παγορευμένα προϊόντα, τόσα προϊόντα απομίμησης, αγορές που ε, έρχονται από δεν ξέρουμε από πού. Βεβαίως μια οδηγία, υπάρχει οδηγία για τις εξαποστάσεως αγορές αλλά ήταν σημαντικό να ανοίξουμε ξανά τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία. Το 2010 ε, ο τζίρος το ήταν 20% παραπάνω. 15 με 17% των καταναλωτών περισσότεροι έγιναν, ε, ε, ε, είναι εξοικειωμένοι με την online αγορά. Για τους καταναλωτές αυτούς πρέπει να δίνουμε νέα πλονεκτήματα. Θεωρώ ότι η οδηγία αυτή προσπαθεί να βελτιώσει την υγιή, τον υγιή ανταγωνισμό και να επιτρέψει τις επιχειρήσεις που ε, να καταλάβουν που αυτή τη στιγμή πουλάνε διαφορετικές, σε διαφορετικές τιμές από τη μία χώρα την άλλη, να το καταλάβουν και να προσφέρουν ανταγωνιστικότερα προϊόντα σε όλους τους καταναλωτές. Αυτό είναι ευκαιρία να, για τον καταναλωτή ότι μπορεί να αγοράζει ανά την Ευρώπη μέσω ίντερνετ. Μεγαλύτερες επιλογές, φτηνότερη τιμή. Το ίδιο ε, θετικό είναι και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες τις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως τις μικρομεσαίες, που έχουν πολύ μικρή γκάμα προϊόντων σε μια κοινωνία που το προϊόντα είναι όλο και πιο εξειδικευμένα το να μπορούν να εκμεταλλευτούν εκατοντάδες ε, εκατομμυρίων καταναλωτών ε, μακριά ενδεχόμενα από το σημείο εγκατάστασή τους είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Ωστόσο και μάλλον και το λέω αυτό ω Ευρωπαίο, για να δουλέψει το σύστημα χρειαζόμαστε και ένα βαθμό εναρμόνισης. Αλλιώς δεν θα λειτουργήσει. Εάν κάθε, αν κάθε επιχείρηση, όπως συμβαίνει τώρα, πρέπει να ξέρει το δίκαιο της καταναλωτικής ε, χρήσης 27 ε, χωρών, αυτό συμβαίνει τώρα, δεν θα γίνει, δεν θα μπορέσει να πουλήσει. Ζητώ λοιπόν από, τις, ε, από τους συναδέλφους του κ. Γκέπχαρτ, χρειαζόμαστε μια κάποια εναρμόνιση. Όχι παντού. Και σε σχέση με τη γενικευμένη, πρόταση, με τη γενικευμένη εναρμόνιση του, του σχεδίου οδηγία έχουμε αλλάξει. Είναι ωστόσο καθοριστικό να υπάρξει ε, μια κάποια εναρμόνιση ιδίως για τις εξαποστάσεως πωλήσει, ε, όπου δεν υπάρχει φυσική σχέση αγοραστού πολιτού και στις πωλήσει πόρτα-πόρτα ή τις πωλήσει off-premises όπως τις λέμε. Όπως ξέρετε η οικοδόμηση της Ευρώπης στηρίζεται στην ικανότητα να τα βρίσκουμε όλοι για συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένους τομείς. το δίλημα της Ευρώπης είναι ότι δεν μπορούμε να μην προχωρούμε επειδή διαφέρει η κατάσταση από χώρα σε χώρα. Και αυτό ανησυχεί τους καταναλωτές, ότι δεν υπάρχουν βήματα μπρος, ότι υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία και ότι αυτό μπορεί να ε, οδηγήσει σε εγκατάλειψη δικαιωμάτων. Ελπίζω ότι αυτό δεν θα συμβαίνει. Και νομίζω ότι πιο σωστό είναι να πούμε ότι η οδηγία αυτή δεν βελτιώνει τα δικαιώματα των καταναλωτών από το να πούμε ότι τα επιδεινώνει. Όντω η οδηγία δεν βελτιώνει τα πάντα. Πιστεύω ωστόσο ότι δεν πιστεύω ωστόσο ότι οδηγεί σε υποχώρηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Συμβάλλει. Συμβάλλει σε όλες τις χώρες που είναι χώρες που μπήκαν πρόσφατα στην Ένωση και που έχουν δίκαιο καταναλωτικής πιστής που δεν έχει φτάσει στο επίπεδο των ε, δίκαιο προστασία των καταναλωτών, συγγνώμη, που δεν έχει φτάσει στο επίπεδο άλλων χωρών. Οι διατάξει που υπήρχαν σε κάποια χώρα που επέτρεπαν φερειπίν ειδική προστασία του καταναλωτή, χάρη στον κύριο Σφάμπε, μπορεί να διατηρηθεί, παραμένει στην σημερινή οδηγία. Ίσως να αμφισβητήσει αυτό που θα πω ο κύριος Χάρμπορ. Το παράδειγμα που αναφέρθηκε, η Υπάρχει προστασία καταναλωτή στη Μεγάλη Βρετανία για την πολύ, για την πολύ μικρών καταναλωτική πίστη. Κάτι. Γιατί λοιπόν να μην ε, παραμείνει κάτι ε, καλύτερης προστασίας του Βρετανού καταναλωτή από αυτό που φέρνει η οδηγία. Τελειώνω. Βρισκόμαστε σε μία καμπή. Μπορούμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, θα προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε έχοντας πάντα υπόψη μας ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ταυτόχρονα και δυναμική της εσωτερικής αγοράς και υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή που πάνε μαζί, δεν είναι κόντρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, θα μιλήσω Δανίσκα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ η σημερινή ψηφοφορία κατέδειξε κάτι και αυτό είναι ότι οι πράσινοι το αποτέλεσμα αυτό δεν μπόρεσαν να το υποστηρίξουν. Και αυτό οφείλεται ουσιαστικά σε, τρεις, σε τρία επιχειρήματα. Πρώτον, επειδή εδώ πρόκειται για ένα υψηλό βαθμό πλήρου εναρμονισμού και αυτό είναι κάτι που πραγματικά αποτελεί επιδείνωση και η Evelyn Γκέπαρτ έδωσε αρκετά παραδείγματα και υπάρχουν και πιο πολλά που μπορούν να παριθμηθούν. Δεύτερος λόγος, Πολύ λίγη πρόοδο σημαίνει αυτό συνεπάγεται για τους καταναλωτές στην Ευρώπη. Consumers Rights uh, Directive, δηλαδή η Οδηγία περί δικαιωμάτων των καταναλωτών. Είχαμε μεγάλες προσδοκίες ότι θα γινόντουσαν νέα βήματα για να διασφαλιστούν νέα δικαιώματα των καταναλωτών. Δεν έγιναν και δεν κατοχυρώνονται από αυτή την οδηγία. Υπήρξε υπερβολικό πηγενέλα ε, διακυμάνσεις στο πολιτικό επίπεδο και πολύ λίγες σαφείς θέσεις και τοποθετήσεις και γι' αυτό ήταν δύσκολο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία εμεί για τον κύριο Σφαμπ και τον κύριο Σβάμπ. Μπορώ να πω ότι ναι, συμμερίζομαι την άποψη ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό για την ενιαία εσωτερική αγορά αν διευρυνθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αληθεύει αυτό. Χρειαζόμαστε κάπω, α το πω έτσι, πληρέστερο πλαίσιο, ένα πληρέστερο πλαίσιο εναρμονισμού. Αν όμω θέλουμε πλήρη εναρμονισμό, τότε πρέπει πραγματικά το περιεχόμενο, η ουσία του κειμένου να μπορεί να βρίσκεται υπό έλεγχο. Η ουσία και το επίπεδο πρέπει να διασφαλιστούν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Δεν το καταφέραμε αυτό, γι' αυτό έπρεπε να καταψηφίσω. Τούτων λεχθέντων όμω, πιστεύω ότι προχωρήσαμε πολύ από κοινού και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω κάποια πράσινα σημεία ως θέσεις πρασίνων έχουν ενταχθεί. Για παράδειγμα, βελτιωμένοι ορισμοί, σε σχέση με τον ορισμό των καταναλωτών. Έχει βελτιωθεί πολύ το πλαίσιο του ορισμού που χρησιμοποιείται για τους καταναλωτές. Υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης και πληροφόρησης για συμβάσεις όσον αφορά τους εμπορικούς χώρους των καταστημάτων. Βελτιώσαμε, είχαμε, καταλήξαμε και επί της ουσίας σε βελτιώσεις. Ένα κατόφλι, ε, threshold, ένα κατόφλι, μπερδεύομαι με την αγγλική ορολογία, αλλά αυτή είναι η ορολογία που χρησιμοποιήσαμε, η αγγλική. Ένα κατόφλι λοιπόν για χαμηλότερο ποσό ευρώ. Όλες οι συμβάσεις πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό ε, καλύπτονται από την ε, οδηγία με αυτόν τον τρόπο. Και στο τέλος τέλος ε, ε, ποιος έχει το βάρος να αποδείξει κάτι, οι πολιτές. Αυτό είναι, αυτά είναι σημεία που καταδεικνύουν το τι έγινε και πρέπει να ευχαριστήσω για τα όσα επετεύχθησαν. Ήταν δυσχερή η πορεία. Πολλά πράγματα υπήρξαν με τα οποία δεν συμφωνούσαμε και ένα επιπλέον σημείο είναι το άρθρο 26 έχει μεγάλο δυναμικό πρέπει να πω. Δυναμικό ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να έχουν ελευθερία επιλογής. Ελευθερία επιλογής όταν υπάρχουν κάποια προβλήματα με το αγαθό, με το εμπόρευμα που αγοράζουν. Όταν χαλάει για παράδειγμα, έχει κάποια βλάβη, πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι αν ή θα το ανταλλάξουν με καινούριο ή θα, διορθωθεί η ζημιά ή θα επιστραφεί το ποσό που έχουν πληρώσει. Αυτό είναι μεγάλη πρόοδος. Είχα γυρίσει σε ένα κατάστημα πριν από κάποιες εβδομάδες και είπα ότι θέλω να το διορθώσετε αυτό. Ε, και τι θα κάνω στο μεσοδιάστημα, δεν μπορούσαν να δώσουν απάντηση. Να μου διέθεταν μια άλλη συσκευή για το, με το μεσοδιάστημα. Αυτά είναι θέματα που για εμά τους πρασίνους είναι σημαντικά. Μέχρι την Ολομέλεια μπορούμε επικοδομητικά νομίζω να συνεχίσουμε την συνεργασία, να επιληθούν αυτό, αυτά. Ωραίο θα ήταν να καταλήγαμε σε μια συμφωνία, αλλά μπορεί να υπάρξει και μια βελτίωση σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων. Σαφή αιτήματα έχουμε ακόμη προ τον εισηγητή και πρέπει να ε, ε, ρυθμιστούν. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ που βρεθήκαμε. Ένα τελευταίο σημείο θα ήθελα να αναφέρω και αυτό είναι το εξή. Προσέξτε, συμβαίνει το εξή. Πρόκειται για τι διαδικασίε, τι διεργασίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τα θεσμικά όργανα. Ε, αισθάνομαι μια πολύ μεγάλη πίεση σε σχέση με μια συμφωνία στην πρώτη κιόλα ανάγνωση με το Συμβούλιο και από κάποιε κυβερνήσει στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό εμεί ω Κοινοβούλιο να καταφέρουμε να προβληματιστούμε όσον αφορά τι δημοκρατικέ διαδικασίε, ποια συνέχεια θα δώσουμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τάση. Μια τάση που τίνει να συμφωνούμε σε πρώτη ανάγνωση. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά όλα τα θέματα. Είναι και ένα αίτημα προ τι κοινοβουλευτικέ ομάδε του Κοινοβουλίου. Πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη. Διότι υπό πίεση δεν θα έπρεπε να συρρυκνωθεί η δημοκρατική διαδικασία. Δεν θα θέλαμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λίγα λόγια στα πρακτικά. Λίγα λόγια στα πρακτικά από μένα ως εκπρόσωπος των Ευρωπαίων, και, Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Δεν ήμουν σχεδόν ηγητές, αλλά θα σας αναπτύξω τη θέση μας. Συμφωνώ με τους συναδέλφους πως όλες οι πολιτικές ομάδες απέρριψαν την αρχική στρατηγική της Κομισιόν περί μέγιστης εναρμόνισης. Αυτό ήταν μέρο του προβλήματος ε, του όλου αυτού κειμένου, γιατί κατ' ουσίαν είχε σχεδιαστεί να κάνει ένα πράγμα και εμείς το προσαρμόσαμε για να κάνει κάτι άλλο. Νομίζω πως οι αιστείες πρέπει να είναι το πώς θα μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε την προσθέμενη αξία προς τους καταναλωτές από τη διαδικασία αυτή, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αυτό το οποίο θεωρούμε αναγκαία απλοποίηση για τις επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν π.χ. τα κενά πληροφορίε με μία ομάδα προτάσεων και να γίνουν τα πράγματα πιο σαφή και πληροφοριακά για τους καταναλωτές. Και νομίζω πως ειδικά στον κόσμο του διαδικτύου και εκεί όπου μιλάμε για πωλήσει πόρτα-πόρτα και εξ αποστάσεως, νομίζω πως θέλουμε να διατηρήσουμε τα δικαιώματα στο μέτρο του δυνατού. Αλλά το σημαντικότερο κατά την άποψή μας είναι πως έχουμε τώρα ένα ενοποιημένο κείμενο. Νομίζω πως ο εισηγητής θα δεχτεί πως χρειάζεται ακόμη περισσότερη δουλειά γιατί οπωσδήποτε με τόσο πολύπλοκο κείμενο θα πρέπει να δούμε ε, κάποιες ε, συνέπειες, ε, κάποιες βελτιώσεις, ε, το που μπορούμε να βρούμε περισσότερη στήριξη για το κείμενο πριν πάει στην Ολομέλεια. Επίσης, η άλλη κριτική που ασκήθηκε από το Κοινοβουλίο προς την Κομισιόν ήταν πως ε, η οδηγία αυτή δεν λάμβανε υπόψη τις μελλοντικέ εξελίξεις, δηλαδή μιλάμε για ψηφιακά προϊόντα. Υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις ε, οι οποίες θα πρέπει ίσως να δοκιμαστούν αλλά πάνω απ' όλα νομίζω πως αυτή είναι η ισορροπία την οποία αναζητούμε. Και απαντώντας σε αυτό το οποίο είπε η ε, υπό την ιδιότητα του Προέδρου τώρα για την επόμενη φάση της διαδικασίας, το κείμενο αυτό είναι στη συναπόφαση, έτσι εργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον νομοθετικό μας ρόλο. Ψηφίσαμε λοιπόν στην Επιτροπή μας και η έκθεση αυτή θα πρέπει να υιοθετηθεί από το σύνολο του Κοινοβουλίου και θα πρέπει μετά να μπούμε σε συζητήσεις με το Συμβούλιο, δηλαδή όλα τα κράτη-μέλη, για να δούμε πώς θα βρούμε ένα συμβιβασμό. Σε ένα κείμενο τόσο πολύπλοκο όσο αυτό, Νομίζω πως ε, θα πρέπει να γίνει αυτό σε δύο αναγνώσεις και υπό εξαιρετικέ συνθήκε νομίζω θα γίνουν κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η φυσιολογική διαδικασία γιατί μετά στη δεύτερη ανάγνωση έχουμε περισσότερο χρόνο να δούμε τις λεπτομέρειες. Αλλά οι συζητήσει αυτέ είναι ακόμα ανοιχτέ και επιτάπητος. Και αυτό θα το κάνει ο Πρόεδρος μαζί με όλες τι πολιτικές ομάδες για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια συμφωνία. Το χειρότερο δυνατόν θα ήταν να υπάρχει τέτοια απόσταση μεταξύ των θέσεων των δικών μας και των κρατών μελών ώστε να πάγωνε η συζήτηση. Αυτό θα ήταν κακό για τους καταναλωτές. Έχουμε αρκετά παράμετρα εδώ πέρα για να επιτευχθεί πρόοδος και ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε. Τελειώνω εδώ πέρα και δεν έχουμε ερωτήσεις, αλλά να πω πως ε, αν είστε δημοσιογράφος έχετε πάρα πολλές πληροφορίες γιατί αύριο θα έχουμε ένα σεμινάριο για το ιστορικό και τις λεπτομέρειες αυτής της σημαντικής πρότασης, ένα εργαστήριο για τους δημοσιογράφους στην αίθουσα 7 σε 50 στο κτίριο Paul Henry Spack ε, περνώντας την Πασαρέλα απέναντι από τις 9 και 4 μέχρι τις 12 και 4 και νομίζω πως ε, και όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα είναι προσκεκλημένοι μαζί με τους άλλους ειδικού. Οπότε, δεν ξέρω τι, ε, υπάρχουν ερωτήσεις. Κοιτώ εδώ πέρα. Υπάρχει κανένας δημοσιογράφος που θέλει να κάνει ερωτήσεις. Ναι, αναφέρατε τα ψηφιακά προϊόντα. Κάνατε προτάσεις για αλλαγές στο κατέβασμα ή τέτοιες ε, ψηφιακές πίσεις. Τζένιφερ Μπέικερ από την IDG. Α, να μιλήσω γερμανικά. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή αξιολογεί την κατάσταση για τις νομικές και υλικές ελλείψεις αλλά και από την άλλη για το δικαίωμα υπαναχώρησης στα ψηφιακά προϊόντα ως Επιτροπή και ως εισηγητής με τους και ε, αναθέσαμε στον καθηγητή Σμιτιές Ελμία μελέτη που μας την παρουσίασε άλλωστε και οι των καταναλωτών έχουν προετοιμάσει μια μελέτη το αποφασιστικό είναι το πώς θα ισχύσουν πλήρως τα δικαιώματα του καταναλωτή αφενός και αφετέρου να προστατευτεί η πνευματική ιδιοκτησία του παραγωγού. Δεν είναι εύκολη αυτή η μέση οδός ε, να βρεθεί. Έχουμε, έχουμε εκείνα τα ψηφιακά προϊόντα τα οποία ε, είναι στη διάθεση του καταναλωτή για διαρκή χρήση, όπως τα ορίζει δηλαδή η οδηγία και βεβαίως όταν χρησιμοποιηθεί το προϊόν αποκλείεται το δικαίωμα υπαναχώρησης. Οπότε η καλύτερη και μόνη λύση θα είναι να συνεχίσουμε να αξιολογούμε, αλλά θέλουμε να ακούσουμε και την άποψη των καταναλωτών για να λάβει υπόψη της και το μέλλον αυτή η οδηγία Δηλαδή, ακόμα και όταν η διαχωριστική γραμμή μεταξύ πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων καταναλωτών είναι πάρα πολύ δύσκολο να οριστεί. Να πω και εγώ κάποια πράγματα, λέει η κυρία Γκέπχαρτ. Πράγματι, συμπεριλαμβάνονται τα ψηφιακά προϊόντα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και είχαμε συμφωνήσει όλοι. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουμε στον τομέα αυτών ορίσαμε ως αγαθό τα ψηφιακά προϊόντα γιατί οι ορισμοί είναι στο άρθρο 11 το οποίο αναφέρεται και περιορίζεται στις υπηρεσίες. Αυτό συμβαίνει παραδείγματος χάρη όταν ένας έμπορος μου δωρίζει διαφημιστικό ένα DVD μετά το χρησιμοποιώ και μετά χωρίς να το ξέρω ε, συνδέεται με αυτό μία υπηρεσία. Τι συμβαίνει τότε, έχω πέσει σε μία παγίδα που θα μου κοστίσει, τι γίνεται. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουν ακόμα, τα οποία θα ήθελα να συζητήσω με τον κύριο Σβά πριν από την Ολομέλεια, έτσι ώστε να έχουμε μία βελτίωση και εδώ πέρα του κειμένου. Να προσθέσω μία πρόταση για αυτό το οποίο είπε ο πτωσναρφός Ρομπέρος Φώ θεωρώ πως ένα από τα λάθη τα οποία γίνεται ξανά και ξανά είναι πως ε, η οδηγία, τέλος πάντων αυτό το οποίο αποφασίσαμε σήμερα, συγκρίνεται με, το, με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι πάρα πολύ κακή. Αυτό το οποίο έκανα εγώ πάντα είναι να τα συγκρίνω με αυτό το οποίο ισχύει σήμερα ως δίκαιο. Όχι πρόταση της Κομισιόν, που ήταν κατά πολύ χειρότερη από το ισχύον δίκαιο στα κράτη-μέλη. Και έτσι συγκρίνω εγώ και αξιολογώ το εάν υπάρχει πράγματι μία ε, προσθέμενη αξία με την ε, οδηγία περί καταναλωτών. Γι' αυτό η απάντησή μου στο τέλος δεν ήταν ναι, εντάξει, είναι σαφώς καλύτερο από αυτό το οποίο πρότεινε η Κομισιόν, αναμφίβολα. Αυτό το είπε και ο κύριος Σφραπ και όλοι βεβαίως ε, και εργαστήκαν πάρα πολύ. Αλλά όχι εάν το συγκρίνουμε με την τρέχουσα κατάσταση στα κράτη-μέλη. Σε κάποιους τομείς είναι επιδείνωση. Και βεβαίως αυτό δεν ε, νομίζω να είναι αποδεκτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα για το θέμα των ψηφιακών προϊόντων. Δεν είναι κάποιο μυστικό ότι δεν είναι καθόλου απλό το θέμα και πρέπει να πούμε ότι τα ψηφιακά αυτά προϊόντα να καλυφθούν από μια οδηγία όπου ουσιαστικά πρόκειται για συγκεκριμένα χειροπιαστά προϊόντα. Είναι τεράστια η πρόκληση για όλο τον ψηφιακό κόσμο. Δεν μπορεί ακριβώς όλα αυτά να ρυθμιστούν ε, όπως ε, σε σχέση με τους φυσικούς νόμους για παράδειγμα ε, με κάποιες διατάξεις. Εδώ προσπαθήσαμε να επιτύχουμε τύχουμε έναν ελάχιστο, ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας καταναλωτών πριν αγοράσει κάποιος μια ταινία, ένα DVD, ένα ψηφιακό τέτοιο αντικείμενο ως υλικό. Και αν κάτι συμβαίνει θα έχει την δυνατότητα να πει δεν λειτουργούσε σωστά και κάτι έχει συμβεί. Όμως αυτό το οποίο δεν είναι εφικτό, δεν είναι δυνατό να γίνει και στο μέλλον θα πρέπει να εξεταστεί είναι το δικαίωμα ανάκλησης ή, ή παναχώρησης. Όταν πατάει κανείς ένα κουμπάκι και έχει το κλικ, ένα κλικ, τότε έχει ήδη κάτι ίσω συμβεί. Όταν φορτώνει κάποιο ή παίρνει κάποιο, κάποιο στοιχεία, αντλεί στοιχεία από τον υπολογιστή, τότε δεν υπάρχει πια δυνατότητα ανάκληση. Πρέπει να δούμε τι είναι εφικτό και τι όχι ψηφιακά. Στο μέλλον θα μάθουμε περισσότερα και θα μπορέσουμε να κάνουμε και περισσότερα. Ευχαριστώ. Άλλε ερωτήσει. Άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ όλους σας που ήσασταν παρόντες, όσους μας βλέπουν ε, ε, στο ίντερνετ. Σας θυμίζω το αυριανό σεμινάριο και ε, αν θέλετε να, να ρωτήσετε τους συναδέλφους κάτι ακόμα, με χαρά να σας απαντήσουν. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε τους διερμηνείς. Καλό σας βράδυ.